Uh, Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας uh, καλωσορίσω θερμά τα μέλη της Επιτροπής, τους καλεσμένους μας για τη δημόσια ακρόαση. Ε, δυστυχώς, uh, λόγω της θέσης μου, δεν βλέπω την ακραριστερά φτέρυγα. Σε λίγο θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους του πάνελ γιατί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ακρόαση επί της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πωλήσεων και μια καλή επιλογή για τους καταναλωτές. Με ερωτηματικό βέβαια, γιατί αυτό θα συζητήσουμε στη δημόσια μας ακρόαση, κατά πόσο θα είναι καλή επιλογή για τους καταναλωτές. Θα ήθελα να κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις ως προς το έργο της Επιτροπής μας για το επόμενο διήμερο. Καταρχήν, η δημόσια πρόσκληση. Γενικώ συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανά. Ελπίζω να μας ακούν πολύ μέσω του διαδικτύου και να μας παρακολουθούν. Τους καλωσορίζω λοιπόν. Επίσης θα γνωρίζετε ότι στην Επιτροπή μας ε, εργαζόμαστε εργοδός για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου το οποίο υπάρχει σε πολλά αντίγραφα και στην αίθουσα αλλά διατίθεται και ηλεκτρονικά με πολλές συνδέσεις ε, που παραπέμπουν και σε άλλα σχετικά έγγραφα. Πολύ ευχαριστώ λοιπόν να σας στείλω και ηλεκτρονικό αντίγραφο και αν δεν έχετε ήδη ενταχθεί στο δίκτυό μας φίλοι της ΙΜΚΟ, της, Επιτροπή, της Επιτροπής μας, ε, σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα μας Εκεί θα βρείτε την σύνδεση και μπορείτε να μας στείλετε ε, το, ενδιαφέρον σας, το ενδιαφέρον για να σας αποστέλουμε την, ε, το ενημερωτικό μας ε, φυλάδιο. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο. Επίσης να εγκρίνουμε και επίσημα την ημερήσια μας διάταξη για το σύνολο της συνεδρίασης. Μέχρι τις 5.30 σήμερα θα παρακολουθήσουμε την ακρόαση για το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο και μετά θα έρθει η κυρία Μπάστος για να μας παρουσιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες ε, για την έκθεσή της που αφορά τους 20 κύριους λόγους ανησυχίας των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Είστε ευπρόσδεκτοι και σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των πολιτών στην ενιαία αγορά. Αύριο επίσημα η συνεδρίασή μας η δημόσια αρχή στις 10 με ώρα ψηφοφορίας και κατόπιν θα έχουμε την πρώτη συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων για την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και καλύτερη διακυβέρνηση ενιαίας αγοράς. Περνάμε τώρα στη δημόσια ακρόαση. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, έγκριτους εμπειρογνώμονές μας. Έχετε λάβει αντίγραφο των βιογραφικών τους. Δεν πρόκειται να κάνω λοιπόν μακροσκελή εισαγωγή. Τους καλωσορίζω θερμά και θα τους δώσω σε λίγο το λόγο. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω το χρόνο αγόρευσης που δικαιούται ο καθένας. 10 λεπτά στον κάθε εμπειρογνώμονα και έχουμε και το πολύ διάσημο μας ρολόι της ΥΜΠΟ. θα το βλέπετε, βλέπετε στις οθόνες για να μην ξεπεράσετε το χρόνο σας και να μπορέσουμε να συζητήσουμε μετά, να έχουμε χρόνο και για τη συζήτηση. Πρώτα θα μιλήσουμε για την παρούσα κατάσταση της, του δικαίου των συμβάσεων με τον καθηγητή Ζουλ Στουκ που είναι διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και του Κέντρου Μελετών ε, Δικαίου του Καταναλωτή στο Πανεπιστήμιο της ε, Λούβεν. Ε, είναι πολύ πεπειραμένος για αυτά τα θέματα και κατόπιν θα περάσουμε στα στοιχεία του κολλήσεων που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μανίκο Γιένς, Γενική Διευθύντρια της ΜΠΕΚ. Θα μας παρουσιάσει τη γνώμη του Γραφείου όλων των οργανώσεων καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα ήθελα να καλασορίσω και πολλούς εκπροσώπους των εθνικών οργανώσεων καταναλωτή. Μου είπαν ότι είναι αρκετοί εκπρόσωποι των καταναλωτών εδώ στην αίθουσα Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε πού κάθεστε, σηκώστε τα χέρια να δω ποιοι είστε. Βλέπω ότι είναι αρκετοί εκπρόσωποι των καταναλωτών, ως ευπαρέστητε. Και φαντάζομαι αργότερα θα επιδιώξετε και επαφή με τους ευρωβουλευτές. Στο δεύτερο τμήμα θα έχουμε λοιπόν την προστασία του καταναλωτή. Μετά από κάθε τμήμα όμως θα προβλέψουμε και ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Και το τρίτο τμήμα αφορά το δικαίωμα υπαναχώρηση από τη Σύμβαση σε σχέση με κάποιες διατάξεις τη οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Εκεί θα έχουμε τον Christopher Warner από την WITCH, που είναι η αρμόδια οργάνωση καταναλωτή του Ηνωμένου Βασιλείου και τον δόκτωρα Ρούπερτ Bellinghaus από την Linklater τη Γερμανία. Και φυσικά ερωταπαντήσει μετά και το τρίτο τμήμα. Πρώτα όμως ήθελα να καλωσορίσω τους δύο αρμόδιους συγγητές μας, την Evelyn Γκέπχαρτ, που είναι γνωστή σε πολλούς από εσά. Ε, είναι και σοσιαλίστρια, συντονίστρια. Χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για μια επέμβαση. Τη ευχόμαστε περαστικά. Ελπίζω να αναρώσει γρήγορα και να είναι πάλι κοντά μας. Μπορεί να μα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Θα την αντικαταστήσει η κυρία Όλγα Σεναλόβα. Έχει Τη ομιλίες τη κυρίας Γκέπχαρτ και θα ακούσουμε και τον Χάν Πίτερ Μάγερ του ΕΛΚ που είναι ο δεύτερος συζητητής, συνεισηγητής με την κυρία Γκέπχαρτ για το θέμα αυτό. Δεν έχω αποφασίσει ποιο θα μιλήσει πρώτο, μια και όμω ο κύριο Χάν Πίτερ Μάγερ είναι ο επίσημο συγγετή. Καλύτερα να μιλήσει πρώτα και να μην έχουμε το ότι προηγούνται οι κυρίε αυτή τη φορά και μετά η κυρία Σεναλόβα ε, σε αναπλήρωση της κυρίας Γκέπχαρτ και κατόπιν θα ακούσουμε τον καθηγητή Ζουλ Στόικ. Κύριε Μάιερ, παρακαλώ, πείτε μας ποια είναι η δική σας προοπτική για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, στην σημερινή η σημερινή ακρόαση θα ασχοληθεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ε, κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων και αυτό είναι το θέμα μας. Είναι προφανές ότι ε, σε σχέση με την πρόταση οι απόψεις μας αποκλίνουν σε ορισμένα σημεία πάρα πολύ και αυτό αναφέρεται τόσο και στις απόψεις των κρατών μελών όσο και των εθνικών κοινοβουλίων και των ενδιαφερομένων συμφερόντων των διαφόρων ευρωβουλευτών, των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε προφανώς, ξέρετε ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ έχει προχωρήσει περισσότερο, διότι η συνάδελφος της ενίδη κατέθεσε τη γνωμοδότησή της με μεγάλη επιτυχία και επικρότηση και τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ αναφερόμαστε εις ε, την ε, εφαρμογή των ε, εταιριών παροχής υπηρεσιών, των ασφαλιών και θέλουμε να καλύψουμε τον καταναλωτή, να τον προστατεύσουμε. Αλλά τονίζω ότι θα θέλαμε να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα ισορροπημένο, μία νομοθεσία η οποία θα είναι ε, ικανοποιητική για όλους και αυτός είναι ο στόχος της προσπάθειάς μας. Δεν θέλουμε απλώς ε, να ε, παρουσιάσουμε μία νομοθεσία που ορισμένοι θα απορρίψουν και δεν θα χρησιμοποιήσουν. Θέλουμε κάτι το οποίο να μπορούμε να βελτιώσουμε, να αμβλύνουμε και ενδεχομένως να το καταστήσουμε πιο πιο ε, σαφές και γι' αυτό περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων αλλά και των ειδικών εμπειρογνωμών που έχουμε καλέξει και ελπίζω να είναι ικανοποιητική η συζήτηση την οποία θα κάνουμε. Ωραία, ευχαριστώ. Η κυρία Σανέλοβα. Και με συγχωρείτε, ο κύριος Στάντεν Μάουιερ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανεφέρθη στην εισαγωγή μου. Είναι ο υπεύθυνο της ε, γενική διεύθυνση που έχει αναλάβει το φάκελο αυτό και ελπίζω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να τον περιλάβουμε ε, στου στους ομιλητές για να μα κάνει ορισμένα σχόλια. Ευχαριστώ η κυρία Σανέλοβα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Χάρμπορ, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι φιλοξενούμενοι, ξέρετε ότι εδώ μιλώ εν ονόματι της κυρίας ε, Γκέπχαρτ η οποία ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί και με παρεκάλεσε να παρουσιάσω τη θέση της σε αυτό το σημαντικό θέμα. Όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο του πολίσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε ε, την ικανοποιητική ελάχιστη προστασία των καταναλωτών που έχουμε θεσπίσει ή θα ζητήσουμε να ευθυγραμμιστούν τα 28 εθνικά δίκαια, πράγμα το οποίο θα δυσχεράνει τη θέση των καταναλωτών διότι η κοινή νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν υπάρχει σωστή προσφορά υπηρεσιών στον καταναλωτή. Όσον αφορά την ε, νομοθεσία ε, της ΡΟΜ 1 εξασφαλίζει στους καταναλωτές ότι πάντοτε θα μπορούν να βασιστούν στην υψηλή προστασία των κρατών μελών τους ακόμη και για διασυνοριακές συναλλαγές. Ενδέχεται κατά το Κοινοβούλιο αυτό να δημιουργήσει ένα προηγούμενο και να οδηγήσει σε μια επέκταση των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε άλλους, ε, σε άλλους τομείς της πολιτικής που αναφέρονται στον καταναλωτή και να μειώσει τα επιτέχματα, τα νομικά που έχουμε επιτύχει για την προστασία του καταναλωτή στην Ευρώπη. Ε, οι συνάδελφοι όμως και ο συνεισηγητής μου πιστεύουν ότι δεν πρέπει να μειωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη παρέχει μία προστασία και θεωρούμε ότι πρόταση αυτή ε, θα βελτιώσει ε, το ε, και που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια αναφερόμαστε στους καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα θέματα του κεκτημένου έχουν εναρμονιστεί μόνο κατά το ελάχιστο και προσφέρουν ελάχιστη προστασία τους πολίτες. Οπότε η πρόταση κοινή νομοθεσίας ως έχει τώρα δεν θα βελτιώσει την κατάσταση αλλά θα οδηγήσει σε μία επιδίνωση της κατάστασης για τους καταναλωτές ορισμένων χωρών. Ε, και γι' αυτό ευχαρίστως θα ακούσω τα σχόλια των εμπειρογνωμών μας επ' και τέλος θα κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι έχοντας μελετήσει τα στοιχεία έχω ερωτηματικά ως προς την ποιότητα και κατακρίνω ιδιαίτερο στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσπάθησε να λάβει υπόψη της την εναρμόνιση ε, ορισμένων θεμάτων ενώ αναφέρεται σε πλήρη εναρμόνιση των ε, υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς ε, τον καταναλωτή. Έτσι όμως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος της συναλλαγής ε, και δεν μπορώ να ακολουθήσω σε αυτό τη λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, όσον αφορά την ανάκτηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών, θεωρώ ότι πρέπει νομοθεσία η οποία θα καταρτιστεί να είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Έχουμε καταρτήσει διάφορα κείμενα σχετικά με το κόστος της παροχής των υπηρεσιών και την προστασία και έχουμε υποβάλει στην ε, Νομική Επιτροπή ορισμένα ερωτήματα για να ελέγξουμε την ποιότητα της πρότασης. Ε, αναμένουμε το αποτέλεσμα και το πόρισμα το Δεκέμβριο και αυτό θα μας ε, διευκρινίσει ορισμένα σημεία. Ευχαριστώ όμως για την συμμετοχή σας και ευχαριστώ που θα μας διευκρινίσετε ορισμένα θέματα. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή και να σας ενημερώσω λίγο για τη διαδικασία και για το κοινό που μας παρακολουθεί. Να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δέσμευση για λεπτομεριακό και σχολαστικό έλεγχο των αντικτύπων της κάθε νομοθετικής πρότασης. Είχαμε μια πολύ ζωή συζήτηση ό,τι αφορά τη μελέτη επιπτώσεων αυτής της πρότασης και οι κύριοι Μάγερ και Σενάλαβα θα υποβάλουν και σχετικές ερωτήσεις και φυσικά ε, ενεπλάξαν στην όλη διαδικασία και οι συνάδελφοι της Νομικής Επιτροπής που είναι η καθήλυνα αρμόδια για το θέμα αυτό, αλλά όπως ξέρετε και η δική μας Επιτροπή ενδιαφέρεται έντονα για το θέμα αυτό, γιατί ε, η προστασία του καταναλωτή εμπίπτει στι αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Θα ακούσουμε τώρα τους εμπειρογνώμονές μας και πρώτα τον καθηγητή Στοικ που θα μας δείξει και διαφάνειες. Έχουν μοιραστεί αντίγραφα. Ε, όσοι είστε πιο πίσω θα μπορείτε να βλέπετε τις μεγάλες οθόνες. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση του καθηγητή Στοίκ και μετά θα του υποβάλουμε και ερωτήσεις. Έχετε περίπου ένα δεκάλεπτο κύριε καθηγητά και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ, παρόλο που δεν είναι η πρώτη μου φορά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όπως δεν βλέπετε ακόμη, ε, μου πρότεινα να αναλύσω την παρούσα κατάσταση του δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνω μια σύγκριση με την τελευταία πρόταση για το για το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Έχουμε δύο ε, λύσεις. Μία είναι η εναρμόνιση κάποιων στοιχείων τουλάχιστον, γιατί έχουμε ε, για τις μεταφορές και τηλεπικοινωνίες κάτι τέτοιο και έχουμε και την πρόταση για ένα προαιρετικό ε, νομοθετικό εργαλείο, κάτι που είναι καινοφανές. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να κοιτάξουμε τη διαφάνεια αυτή και να ρίξουμε μία σύντομη ματιά στο κοινοτικό κεκτημένο για τον καταναλωτή. Αρκετά εντυπωσιακό. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω όλα αυτά. Θα σας δώσω απλώς ένα κατάλογο που ξεκίνησε το 1985 με τις συμβάσεις ε, εκτός εμπορικού καταστήματος. Στη συνέχεια έχουμε το πακέτο για την καταναλωτική πίστη, για το πακέτο ταξιδιωτικό, πολύ σημαντικές ε, οδηγίες, γιατί πρόκειται για οριζόντιες οδηγίες που ισχύουν για όλες τις συμβάσεις. Είχαμε το time sharing, τη χρονομίσθωση, συμβάσει εξ αποστάσεως, ε, πολύ πιο ε, ειδικά νομοθετήματα. Επίσης έχουμε τις ε, πωλήσει καταναλωτών, κάπως παραπλανητική αυτή η διατύπωση, γιατί μιλάει μόνο για τη συμμόρφωση, την διετή εγγύηση και εμείς έχουμε την εξαποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μετά στα, στις μεταφορές έχουμε πολλούς κανονισμούς για τις καθυστερήσεις, για άρνηση επιβίβασης, Έχουμε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πολύ σημαντικά μέτρα προστασίας του καταναλωτή στο πακέτο του 2009 και την οδηγία για τις οικουμενικές υπηρεσίες 2009-136 ε, και την περσινή οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή που περιλαμβάνει νέα μέτρα και μερικά μάλιστα ε, τροποποιούν υπάρχοντες κανόνες ενώ μερικά είναι καινούργια. Έχουμε νέους κανόνες για παράδειγμα για τέλη που καταβάλλονται σε περίπτωση χρήσης ε, μέσων ε, πληρωμής, ε, τέλη για επικοινωνία τηλεφωνική και επιπλέον επιπρόσθετες πληρωμές. Επίσης, έχουμε στην οδηγία για την κεφαλαϊκή επάρκεια έχουμε το θέμα της παράδοσης και της μετάθεσης κινδύνου στις πωλήσει σε καταναλωτή. Αυτό το συγκρίνουμε ιδιαίτερα με το προτινόμενο προαιρετικό ε, κοινό ε, ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Τώρα έχουμε εδώ μια σύγκριση μεταξύ του κοινοτικού κεκτημένου, δηλαδή του κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι συμβαλόμενοι δεν έχουν επιλέξει το προαιρετικό αυτό ΚΕΔΠ, το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολίσεων, που παρουσιάζεται ως δεύτερο νομικό καθεστώς εντός του κάθε κράτους μέλους ε, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. Βέβαια το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ισχύει, αλλά εδώ έχουμε ένα δεύτερο νομοθετικό πλέγμα εντός μιας εθνικής νομοθεσίας. Το πεδίο εφαρμογή μόνο συμβάσει πωλήσεων, πωλήσει ψηφιακού περιεχομένου, προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και τέλο ε, ε, συμβάσεις για παροχή συναφών ε, υπηρεσιών, που σχετίζονται δηλαδή με την πώληση αγαθών ή την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου και δεν αφορούν άλλες υπηρεσίες. Δεν αφορά μόνο ε, συμβάσεις επιχειρήσεων με καταναλωτές, όπως το κοινοκτικό κεκτημένο, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων. Αρκεί ένα συμβαλόμενο είναι μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά τα κράτη-μέλη μπορούν να επεκτείνουν την ισχύ και στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, χωρίς να είναι κατά επιχείρηση μικρομεσαία. Ισχύει μόνο για διασυνοριακέ καταστάσει, καταρχήν, μόνο για διασυνοριακέ συμβάσει, αλλά και πάλι τα κράτη-μέλη μπορούν να επεκτείνουν τη χρήση του ΚΕΔΠ και σε εγχώριε συμβάσει. Στο κοινοτικό κεκτημένο έχουμε κανόνε που ε, εφαρμόζονται άσχετα αν υπάρχει ένα διασυνοριακό στοιχείο. Ήδη αναφέρθηκε ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο είναι προαιρετικό, θα πρέπει να συμφωνούν οι συμβαλόμενοι και μάλιστα ε, δεν έχουμε από το κοινωνικό κεκτημένο που επιλέγουν οι επιχειρήσεις και πρέπει απλώς να συνενέσει ο καταναλωτής. Είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διαφορετική τελικά λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ του κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου Πολίσεων και του κοινοτικού κεκτημένου 2, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στι περιπτώσει σύμβαση επιχείρηση και καταναλωτή δεν υπάρχει επιλεκτική εφαρμογή του ΚΕΔ. θα πρέπει κανεί να το εφαρμόσει ολόκληρο ή καθόλου. Δεν μπορεί να επιλέξει μερικέ μόνο διατάξει του. Σημαντικό στοιχείο προστασία του καταναλωτή. Τώρα, ε, μερικές συμβάσεις εκπίπτουν το πεδίο εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου πολίσεων. Για παράδειγμα, ε, νομική προσωπικότητα, παρανομία, ανηθικότητα, γνώση, μη διακριτική μεταχείριση. Στο κοινοτικό κεκτημένο έχουμε πολύ περισσότερα ε, στοιχεία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή. Γιατί εδώ έχουμε μια πολύ, ε, ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα διατάξεων και εδώ έχουμε φυσικά B2B ε, μεταξύ επιχειρήσεων, αρκεί μια επιχείρηση να είναι ε, μικρομεσαία. Επίση, το κοινοτικό και εκτιμένο δεν περιορίζεται σε υπηρεσίε, σε πωλήσει, συγγνώμη, αλλά και σε υπηρεσίε. Ενώ το ΣΕΖΕΛ, το ΚΕΒΠ είναι πιο περιορισμένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει μικρότερη προστασία, ε, υποβαθμισμένη προστασία στου καταναλωτέ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του ΚΕΔΠΑ, τα, τα, οι συμβαλόμενοι ε, εφαρμόζονται de facto μάλλον το κοινοτικό κεκτημένο. Τώρα, μερικές, ε, μερικά πλεονεκτήματα του κοινοευρωπαϊκού δικαίου πολίσεων. Πολύ σημαντικά στοιχεία των πωλήσεων καλύπτονται όπως η σύναψη της σύμβασης, ε, ε, ελαττώματα της ε, βούλησης, ερμηνεία, ένομα βοηθήματα, αποζημιώσεις, τόκοι, περιμερίες, μεταγραφή, απόδοση και το καθεξής. Επίσης υπάρχει μια, ένα σημείωμα, τυποποιημένο σημείωμα ενημερωτικό που εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση Στου καταναλωτέ και φυσικά είναι ο προαιρετικός χαρακτήρας. Απαιτείται ε, να γίνει επιλογή, ρητή επιλογή από τα συμβαλώμενα μέρη. Έκανα συγκρίσεις ε, μεταξύ του νομικού συστήματος ε, του Βελγίου και διαπιστώνω ότι κατά το 90% οι κανόνες του, κοινωνικού, του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του ευρωπαϊκού, του βελγικού δικαίου. Και το ίδιο με, μου είπε και συνάδελφοι από άλλα κράτη-μέλη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το ΚΕΔ θα υποβαθμίσει την προστασία είτε την, ε, την νομική, την εθνική, είτε του κοινοτικού κεκτημένου. Τώρα, για τους αθέμετους όρους, καταχρηστικού όρου. Η οδηγία περιλαμβάνει μια γενική ρήτρα και ένα αναδεικτικό κατάλογο των αθέμητων καταχρηστικών όρων, Πολύ νομολογία σχετική που είναι φιλική προς τον καταναλωτή, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι περίτη εφόσον ε, εγκριθεί το, το το ΚΕΔ. Επίσης, ε, στο Βέλγιο θα ισχύει για τους υποδιαπραγμάτευση όρους. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια, γιατί όλοι οι όροι μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οπότε είναι μάλλον θεωρητικό αυτό το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Δεν υπάρχει γενικό γενική υποχρέωση διαφάνεια με βάση την οδηγία αυτή και έχουμε ένα απλώ ενδεικτικό κατάλογο. Ενώ στο ΚΕΔ έγινε προσπάθεια για να συνταχθεί ένα μαύρο μαύρος μια μαύρη λίστα και ένα μακροσκελή γκρι κατάλογος που εξασφαλίζει μεγαλύτερη βεβαιότητα για του καταναλωτέ. Ένα άλλο παράδειγμα εδώ είναι τα ένομα βοηθήματα του αγοραστή. Γιατί αν ρίξουμε μια ματιά στην οδηγία για τις πωλήσει έχουμε πολλές, πολλά ένομα βοηθήματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αλλά υπάρχει δυνατότητα για τις επιχειρήσεις ε, ε, ε, να προτείνουν επιδιόρθωση και σε περίπτωση που δεν ισχύσει η επιδιόρθωση τότε μπορούν να ζητήσουν καταγγελία της σύμβασης. Το ΚΕΔΠ όμως περιλαμβάνει πολύ περισσότερα ένομα βοηθήματα. Στο 106 έχει το δικαίωμα ε, ε, να ανασταλεί η εκτέλεση, υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης, δεν υπάρχει δικαίωμα ε, διόρθωσης. Οπότε στο ΚΕΔ περιλαμβάνει υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή από το κοινοτικό κεκτημένο. Τώρα, τα υπέρ και τα κατά των δύο καθεστώτων. Φυσικά υπάρχουν και για τις δύο πλευρές ευρύτερο πεδίο εφαρμογή για το ΚΕΖΛ. Τώρα έχουμε ε, για την ομολογία περισσότερο, περισσότερη ομολογία για το κοινοτικό κεκτημένο, για το ΚΕΔ θα πρέπει να περιμένουμε. Επίση, ορισμένα θέματα του κοινοτικού κεκτημένου δεν εμπίπτουν αυτόματα στο κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο πωλήσεων. Και τέλο, εδώ έχουμε νέα σημεία με τι καταληκτικέ μου παρατηρήσει. Δυστυχώ πρέπει να μου δείξετε εδώ εμπιστοσύνη γιατί δεν μπορείτε να ελέγξετε αυτά που λέω. Ορισμένες, μόνο ορισμένα τμήματα του συμβατικού δικαίου των καταναλωτών εναρμονίζονται. Ορισμένες πτυχές όπως η αθέμητη όρη εξαποστάσεως πωλήσει και επίσης έχουμε ειδικού κανόνες για ορισμένες μόνο ε, υπηρεσίες για τις χρηματοπιστωτικές, χρονομίστοση και ταξίδι και όχι για όλες τις ε, υπηρεσίες, αλλά ούτε και στο ΚΕΔΙΠ υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα, το κοινοτικό κεκτημένο είναι ένα μείγμα ελάχιστης και πλήρους εναρμόνη. κάτι που είναι κάπως ε, ε, δημιουργεί σύγχυση, αλλά ίσως είναι και αναπόφευκτο. Τώρα, το σύστημα ενόμων βοηθημάτων στο κοινοτικό κεκτημένο είναι ε, ατελές και από αυτή την άποψη το κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο συνιστά μια βελτίωση. Υπάρχει όμως ε, μέσω των, κανονισμών ε, μία διείσδυση των εθνικών συμβάσεων για τις μεταφορές, ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες. Βέβαια δεν είναι οδηγίες αυτές που μπορεί κανείς ε, να τις εφαρμόσει. Είναι κανονισμοί που υποχρεωτικά εφαρμόζονται. Επίσης υπάρχει ένας κατακαιρματισμός που δημιουργεί κάποια αβεβαιότητα, έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Η διευρύνεται ο ρόλος του ΔΕΚ, που βέβαια είναι πολύ πιο φιλικό Προ το καταναλωτή. Και έτσι ίσως έχουμε πολλή νομολογία, όχι μόνο για το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολίσεων, αλλά και για τις αθέμετες εμπορικέ πρακτικές. Και τέλος, το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων έχει υψηλό επίπεδο προστασία του καταναλωτή, ίσως αποτελέσει ένα επόμενο βήμα στη βελτίωση της προστασία του καταναλωτή στην Ευρώπη. Αυτά και σα ευχαριστώ. Well, thank you. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε που είναι πληρέστατα, πραγματικά. Πράγματι τώρα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα είχαμε προβλέψει ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Οπότε για να δούμε μήπως οι συγητές, η... η κυρία που έχει αναλάβει καθήκοντα συγητή, οι υπόλοιποι που είναι εδώ Α, η κυρία Ρούλε και άλλοι έχουν ζητήσει είναι εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις προς τον καθηγητή Στακ τώρα, πριν να συνεχίσουμε. Κύριε Σβάπ, εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω βέβαια εγώ να αλλάξω τη σειρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, επειδή είπε ο εισηγητής ότι σε σχέση με το βελγικό δίκαιο δεν υπάρχει μία επιδίνωση της θέσεως του καταναλωτή θα ήθελα να ρωτήσω επειδή αντιμετώπισα τις δυσκολίες αυτούς και η αξιολόγηση της ε, συναδέλφου Σενάλοβα την οποία εκτιμώ πάρα πολύ αλλά με την οποία δεν συμφωνώ όσον αφορά τα σχόλια που μας έκανε θα ήθελα να ε, σας πω ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι το επίπεδο της προστασίας καταναλωτών του ΣΕΣΔΙ είναι χαμηλότερο από το επιζητούμενος. Ε, ευχαριστώ. Ε, δεν κατάλαβα. Είπατε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ε, θα συμφωνούσαν ότι υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτό που δεν κατάλαβα όμως ήταν η πλειοψηφία των συμμετεχόντων που από αυτών που εξετάζουν αυτή την οδηγία. Δηλαδή οι περισσότεροι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιζητούμενη προστασία καταναλωτών. Δεν ξέρω πώς ε, υπολογίζεται την πλειοψηφία, ίσως όχι όπως το Κοινοβούλιο, αλλά από τις αντιδράσεις στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων μπορώ να σας πω ε, ε, αξιολογώντας το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε και φτάνοντας στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα ότι εντός της ομάδας μας οι περισσότεροι θα κατέληγαν στην αντίθετη άποψη από την πλειοψηφία της δικιάς σας ομάδας όποια και να είναι αυτή. Είναι μια πολύ ενηγματική προοπτική αυτή κύριε Σβάμπ νομίζω αλλά σαν πρόεδρος θα ήθελα να βασιστώ σε αυτό το επιχείρημα που θέσατε και που είναι ενδιαφέρον διότι τονίζετε ότι η νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν 28ο σύστημα καθεστώς θα προσφέρει μια καλύτερη προστασία των καταναλωτών σε όλους τους τομείς αλλά είναι ένα μέρος της συνολικής προστασίας. Το ερώτημα είναι λοιπόν πού προσφέρει ε, προστιθέμενη αξία το ΣΕΖΛ που όντως αναβαθμίζει την συνολική προστασία και που συμπληρώνει άλλα θέματα τα οποία τονίσατε στην εξαιρετική σας και λεπτομερέστατη ανάλυση. Ε, δηλαδή, εάν κάποιος επιλέξει να ισχύσει το CSSL, ε, τι εναλλακτικές θα έχει για την προστασία του. Είναι ένα περίπλοκο θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς. Γι' αυτό και ο κύριος Φαμπ δήλωσε ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Θα ήθελα να μου πείτε εάν κατάλαβα την ανάλυση σας σωστά και σε περίπτωση όπου όντω έτσι είναι, εάν η προστασία του καταναλωτή πρέπει να είναι 100%, τι ποσοστό αυτής της προστασίας θα μπορέσει να καταλογιστεί ε, σε αυτό το νέο μέσο σε σχέση με άλλα. Θα έλεγα ότι αναφερόμαστε μόνο στις πωλήσει και αυτό υπό την ε, προϋπόθεση ότι οι συμβαλόμενοι θα έχουν επιλέξει το σύστημα αυτό. Δηλαδή έχει σημασία εάν ε, ε, επιλεγεί το σύστημα αυτό ο καταναλωτής θα είναι προστατευμένος. Υπάρχει βέβαια πάντοτε ε, και η εναλλακτική του κεκτημένου της προστασίας του καταναλωτή σε εθνικό επίπεδο και ποιες είναι οι λύσεις σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι. Κύριε Μάγια, θέλετε να σχολιάσετε εσείς. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι το 1985 ε, άρχισαν τα πρώτα ευρωπαϊκά νομοθετήματα για την προστασία του καταναλωτού τα οποία προχώρησαν. Ποια είναι όμως τώρα αυτή η επίπτωση. Εάν ισχύσει αυτή η νέα νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και το δίκαιο των πολίσεων οι περισσότερες από αυτές τις νομοθεσίες θα αρθούν ή θα ε, συνεπάρχουν υπάρχουν και θα έχουν συνοπτιστεί σε ένα συνοπτικό νέο νομοθέτημα. Νομίζω. Νομίζω ότι εδώ παρεύουμε διαφορετικά ζητήματα. Το CSL, το CEDC δηλαδή, θα αφορά ορισμένες συμβάσεις, όχι ταξιδιωτικά πακέτα για παράδειγμα και τέτοια θέματα, τα οποία έχουν ε, τις δικές τους οδηγίες που έχουν λόγω ύπαρξης. Αν ε, βέβαια έχετε συμβάσεις πωλήσεων εξ για παράδειγμα, ή που έρχονται στο σπίτι πολιτές ή στα καταστήματα, τότε οι οδηγίες αυτές για τις συμβάσεις εκείνες που έχει διαλέξει κανείς ε, το νέο σύστημα, ισχύει το νέο σύστημα. Το παλιό βέβαια θα έχει τη δικιά του λειτουργία όσο είναι σε θελοντική βάση το νέο σύστημα. Θα παραμείνει και θα έχει τη λειτουργία που έχει και τώρα. Οπότε, αν επιλέξει κανείς το νέο καθεστώς, θα είναι σε χειρότερη θέση ο καταναλωτής. Αυτό είναι το ερώτημα νομίζω που τίθεται σήμερα. Και απάντησή σήμερα είναι όχι, δεν θα είναι σε χειρότερη θέση. Αλλά εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του άποψη εδώ. Πρόεδρος. Νομίζω πολύ καλά μας θέσατε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η συζήτησή μας σήμερα. Ιδιαίτερα για την προστασία του καταναλωτού και για τα δικαιώματα υπαναχώρησης που θα συζητήσουμε αργότερα. Κανένας άλλος έχει ερωτήσεις? Συνήθως οι βουλευτές ρωτάνε στι ακρόασει. Αλλά παρόλα αυτά, αν από το κοινό που βρίσκεται εδώ, αν κάποιο καίγεται να υποβάλει μια ερώτηση, μπορεί να μου στείλει ένα σημειωματάκι και θα δω αν υπάρχει χρόνο θα αντιθέσουμε την ερώτησή σα. Αλλιώ θα συνεχίσουμε ω ήθιστε. Αλλά σα λέω ότι αν καίγεστε να ρωτήσετε κάτι, ενημερώστε με. Θα προσπαθήσουμε έτσι να καλύψουμε όλα τα θέματα. Τώρα προτείνω να συνεχίσουμε και να περάσουμε στο επόμενο τμήμα που είναι να δούμε τις διάφορες προοπτικές που τίθενται όσον αφορά την προστασία των ε, καταναλωτών από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Έχουμε την κυρία και τον κύριο Σάιφερτ. Είναι κάποιος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα τα παρακολουθεί από το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Είναι και νομικός και μόνιμο μέλος της ομάδας εργασίας για το καταναλωτικό δίκαιο. Θα σας δώσω 10 λεπτά στον καθένα και μετά πάλι θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Και λέω στους εμπειρογνώμονες ότι εννοείται πως στο τέλος της ακρόασης αυτής θα σας δώσω το λόγο για να μας πείτε τη γνώμη σας για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν στο μεταξύ κατά τη διάρκεια της συζήτησης θέλετε να πείτε κάτι, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα η κυρία Γκόγες, λοιπόν, που είναι ε, διευθύντρια του ΜΠΕΚ, που είναι ο Οργανισμός για την Προστασία των Καταναλωτών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και πολύ χαίρομαι που η Επιτροπή σας έχει οργανώσει αυτή την ακρόαση γιατί αυτά τα ζητήματα το κατά πόσο δηλαδή το νέο αυτό προτινόμενο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων είναι μια καλή ιδέα για το καταναλωτή, όχι, επιτέλους πρέπει να συζητηθεί. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας τι σκέψεις μας και τι αναλύσει μα. Πρόεδρε, όπως είπατε, υπάρχουν εδώ στην αίθουσα πάρα πολλέ οργανώσει καταναλωτών. Και γιατί, ακριβώ γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Πολλά έχουμε να πούμε, ξέρω ότι μου δώσατε μόνο 10 λεπτά, οπότε αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες κοιτάξτε την ιστοσελίδα μας ή να συζητήσουμε διμερώς αν θέλετε για αυτά αργότερα. Λοιπόν, από πλευρά του καταναλωτή, όταν μιλάμε για το κέρδομα πρέπει να ρωτηθούμε τρία πράγματα. Πρώτον, οι καταναλωτές χρειάζονται ένα σε θελοντική βάση δίκαιο πολίσεων. Έπειτα, ποιε θα είναι οι επιπτώσει του προτενούμενου συστήματο στον καταναλωτή και τρίτον, ποιε θα είναι οι επιπτώσει του προτενούμενου συστήματο στο μέλλον τη ευρωπαϊκή πολιτική για τον καταναλωτή και τη σχετική νομοθεσία. Να ξέχασα να ξεκινήσω με τις διαφάνειές μου. Να, τώρα θα τις δείτε, λέω Μιλήτρια. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα ε, στέρεο ε, πλαίσιο το οποίο να προστατεύει τους καταναλωτές. Είχαμε την οδηγία του 2011 για την προστασία των καταναλωτών που προβλέπει εναρμόνιση στα πιο σημαντικά σημεία στα αγαθά που πολλούνται online για παράδειγμα. Και το Κοινοβούλιο βοήθησε πάρα πολύ με την νομοθεσία αυτή. Αυτή είναι η επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια μεγάλη αλλαγή στην προσέγγιση της και προτείνει σε θελοντική βάση να υπάρχει ένα μέσο. Αλλά αυτή, αυτό είναι ένα αριθμιστικό θα έλεγα, πείραμα, το οποίο ελοχεύει πολλούς κινδύνους. Έχω ετοιμάσει για την μελέτη αξιολόγησης μια διαφάνεια, αλλά άκουσα ότι έχει συμφωνηθεί ήδη να γίνει, ο δηλαδή έχει συμφωνήσει να γίνει ένας τέτοιος έλεγχος αλλά θα συνοψίσω τη θέση μας ως εξή. Οι οργανώσεις των καταναλωτών και η δικιά μας όλος ιδιαίτερος δεν στηρίζουμε αυτή την πρόταση για κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων. Δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα τέτοιο μέσο. Και ιστορικά μιλώντας είναι μια μοναδική περίπτωση. Εμείς, ο οργανισμός μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο οι οργανώσεις μέλη μας, θέλουν να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν με τις άλλες πλευρές και το έχουν κάνει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό και όλοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί γι' αυτό το νέο μέσο την πρόταση. Αν λοιπόν και ο επιχειρηματικός κόσμος και οι καταναλωτές αμφισβητούν την ε, ανάγκη και το κατά πόσο είναι επιθυμητό ένα τέτοιο σύστημα, γιατί να το κάνουμε. Έπειτα δεν απλοποιείται η ζωή του κόσμου, αντίθετα γίνεται πιο περίπλοκη τόσο των καταναλωτών όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν εξυπηρετούνται οι καταναλωτές, αντίθετα εξυπηρετούνται λιγότερο από ό,τι κατά το παρελθόν και διαφωνώ με τον προλαλήσαντα διότι υπάρχει νομοθεσία για πάρα πολλού ε, τομεί και πριν από το ΚΕΔΜ και εξάλλου μπλοκάρει βελτιώσει ή συγχρονισμό του δικαίου για τους καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι δεν είναι μια καλή προσπάθεια νομοθεσίας, δεν είναι ο σωστός τρόπος να δούμε τις ε, συμβάσεις πωλήσεων. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα δίδυμο νομοθεσίας, δεν αντικαθιστά κάτι, θα υπάρχουν 27 εθνικές νομοθεσίες των χωρών μελών, θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ισχύει και επιπλέον θα υπάρχει και το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Οι ακαδημαϊκοί ειδικοί το λένε ότι είναι περίπλοκο κάτι τέτοιο. Για τους ίδιους, φανταστείτε τι γίνεται για τον απλό κόσμο. Τα δικαστήριά μας πώς θα αντιμετωπίσουν ε, τις περιπτώσεις που θα προκύψουν όταν υπάρχει αντίφαση. Οι νομοθετικές αλλαγές ε, πώς θα εξεταστούν ε, χωριστά, από κοινού, με ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα, εννοείται ότι θα υπάρξουν φυσικά και ένα τσουνάμι ε, προδικαστικά ερωτήματα που θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και θα οδηγηθούμε και σε διακρίσει. γιατί τελικά οι καταναλωτέ ε, θα τυχαίνουν διαφορετική ε, εξεργασία, θα του συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με το αν έχουν διαλέξει το ένα ή το άλλο σύστημα. Οι μεγάλε επιχειρήσει, μην ξεχνάτε, θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα μέσα από αυτό το πολύπλοκο τοπίο, ενώ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν θα τα καταφέρουν. Αλλά διάκριση και στον επιχειρηματικό κόσμο. Εμείς διαφωνούμε και στο εθελοντικό, διότι δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα έτσι, διότι υπάρχουν ζητήματα και στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στο clouding. Δεν ξέρουμε λοιπόν στην εφαρμογή πώς θα λειτουργήσει. Το επίπεδο πάντως της προστασίας των καταναλωτών έτσι όπως προτείνεται ε, στο κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων δεν είναι αρκετά υψηλό όπως ήταν μέχρι τώρα. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, πάντως έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο που έχουμε ετοιμάσει με τη συνεργασία των μελών μας και έχουμε αναλύσει κάθε διάταξη χωριστά. Και σε πολλά σημεία η προστασία που προσφέρεται με αυτό το μέσο είναι χαμηλότερη από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δεν πρέπει λοιπόν να παρασύρουμε τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες να πάρουν σαν μέτρο την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά την εθνική νομοθεσία. Γιατί επ' αυτού πρόκειται, με αυτό πρέπει να συγκρίνει το νέο, την νέα πρόταση ο καταναλωτής. Επαναλαμβάνω ότι για τους καταναλωτές δεν υπάρχει επιλογή. Τους λέμε ή το διαλέγετε ή δεν έχετε τίποτα. Δεν υπάρχει περιθώριο να διαπραγματευτεί δηλαδή ο καταναλωτής για αυτό το νέο μέσο. Από πλευρά λοιπόν πολιτικής είναι πολύ ανησυχητικό το ΚΕΔΠ επίση θα περιορίσει τις εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων που υπάρχουν μέχρι τώρα. Α δούμε το ψηφιακό περιεχόμενο για παράδειγμα. Η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προβλήματος εδώ, γιατί δεν έχουμε προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες. Συνεπώς πρέπει η νομοθεσία να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Εντάξει, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων υποτίθεται ότι το κάνει. Συγχρόνω όμω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πέρα από το κέρδο δεν θέλει καμία νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή ο καταναλωτή να <clears throat> από νέου κανόνε όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο μόνο εφόσον ο ίδιο ο έμπορο αποφασίσει να επιλέξει το αντίστοιχο μέσον. Για μας δεν είναι μια καλή ιδέα αυτό, δεν είναι καλός τρόπος να νομοθετούμε. Τι προτείνουμε, Προτείνουμε να ψάξουμε να βρούμε πρακτικές λύσεις. Προτείνουμε δηλαδή να δουλέψουμε πάνω σε ένα ευρωπαϊκό ε, μοντέλο συμβάσεων που θα καλύπτει τις πωλήσει που γίνονται online μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε μία ε, προσέγγιση soft law, μη υποχρεωτικής ε, δηλαδή και δεσμευτικής ρύθμισης και γρήγορες λύσεις με το ADR-ODR. Θέλουμε κάτι το οποίο εγκρίνουν οι οργανώσεις και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και να μην αντικαθιστά την εθνική νομοθεσία, αλλά να γίνεται διαπραγμάτευση στο υψηλότερο δυνατόν προστασία του καταναλωτών, οπότε οι καταναλωτέ θα έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό, αφού θα το έχουν διαπραγματευτεί προηγουμένω, και θα έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό και οι έμποροι, γιατί θα νιώθουν βεβαιότητα, γιατί θα ξέρουν ότι έχει περάσει από διαπραγμάτευση και άρα ο κίνδυνο θα είναι πολύ μικρό τέτοιε συμβάσει να ε, καταλήξουν κάποια στιγμή στα δικαστήρια, να προσφύγει κάποιο δηλαδή εναντίον του. Εμεί, Έχουμε τέτοιες προτάσεις και τις επεξεργαζόμαστε παρετέρω. Τέλος, πιστεύουμε ότι όντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την ομοθεσία για τις ε, συμβάσεις και για τους καταναλωτές. Όντως υπάρχει θέμα διασυνοριακού εμπορίου, το έχει πει και η Επιτροπή, αλλά το λέει και η δικιά σας ε, η έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει, να λειτουργήσουμε έξυπνα, να ξεπεράσουμε τους ε, φόβους που έχουμε με πρόσβαση στο ADR και στο ODR και να έχουμε μοντέλα σύγχρονων συμβάσεων. Με τον καθηγητή Στέφ συμφωνώ για το ότι υπάρχουν αδυναμίες στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Όντω, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών να εξυγχρονιστούν περισσότερο, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με νομοθεσία από την οποία έχουν αποφεληθεί όλοι οι καταναλωτέ και όχι μόνο εκείνοι που έχουν επιλέξει σε εθελοντική βάση ένα μέσο. Δεν θα πρέπει να είναι εθελοντικό το μέσο, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή να μην υπάρχει. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι για να λειτουργήσει καλά μια αγορά χρειάζεται να κινητοποιούνται οι έμποροι και να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές. Χρειάζονται δίκες συμβάσεις. Δεν είναι δυνατόν αλλιώ να λειτουργήσει μια αγορά. Γι' αυτό και εσείς θα πρέπει να ακούσετε τα ενδιαφερόμενα μέρη και ελπίζω ότι αυτό επιτέλους θα γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις διαφανειές σας. Ήταν πολύ ξεκάθαρες. Όντως τίθονται διάφορα ζητήματα εδώ, τα οποία και θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Ε, ο κύριος Σάιφερ τώρα, που σας είπα, ότι είναι, που είναι από το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, Γερμανία, να μας πει κατά πόσο θεωρεί πως το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων είναι μια καλή ιδέα ή όχι για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να έρχομαι πολύ κοντά στο μικρόφωνο. Ότι μας κυρίες και κύριοι, ε, ο, καθ, ε, προσανατολίστηκα βάσει του τίτλου αυτής της ακροάσεως για ορισμένα στοιχεία και όπως είπε και η κυρία Γκόγενς πρέπει κανείς να αναρωτηθεί αν μπορεί να βρεθεί μία ιδεώδης λύση διότι εμείς στην Γερμανία από το ε, επαγγελματικό επιμελητήριο και εμπορικό επιμελητήριο θεωρούμε ότι ε, ενδέχεται βέβαια να προκύψουν προβλήματα πρέπει να συζητήσουμε αλλά δεν είναι κακή αυτή η ιδέα ε, και τώρα θα ήθελα το πρώτο, την πρώτη σελίδα από τις ε, θεωρώ ότι είναι καλό να μην το ε, επιθυμούμε μόνο εμείς αλλά θα πρέπει να το αποδεχθεί και ο, ο, ο συμβαλόμενος διότι εάν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο των πωλήσεων και των αγορών το οποίο θα ενοποιηθεί διότι διαφορετικά δεν θα το δεχθούν οι έμποροι και οι εμπορικές εταιρείες και επίσης κάτι άλλο το που έχει λεχθεί πολλές φορές το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο προκύπτει σε πολλές συζητήσεις. Επ' αυτού μπορούμε να πούμε μόνο μία λέξη ότι δεν έχουν θέση εδώ και μόνο θα, θα μας συμπαρασύρουν σε προβληματικούς τομείς που δεν χρειαζόμαστε γι' αυτό και συμφωνώ με όλους όσους ε, επενέβησαν σήμερα και είπαν ότι το ψηφιακό περιεχόμενο δεν έχει θέση σε αυτή τη ρύθμιση. Επίσης, όπως είπαμε επανειλημμένως, η αποδοχή ενός τέτοιου προγράμματος σαν το CESL ε, μπορεί να υπάρξει αν υπάρχει μία σταθερή ε, νομική βάση. Πάντοτε λέγεται ε, και αναφέρεται το άρθρο 114 κατά τη γνώμη μας δεν είναι το σωστό και όπως και το 2006 ενδέχεται κάποια μέρα να έρθει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πει ε, ωραία ε, η νομοθεσία σας αλλά δεν έχει νομισή ε, βάση όπως έγινε το 2006 για τις Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Η, η κατάσταση δεν είναι ακριβώς η ίδια αλλά για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Πιο συγκεκριμένα ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς ξεκινούν με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και ε, αυτό βλέπουμε ότι εάν μετρήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται ε, στο ε, ΣΥΣΛ αναφέρονται 97 στο κείμενο και 12 για την πώληση των αγαθών στο διαδίκτυο. Ίσως ε, είμαι προκλητικό στη διατύπωσή μου, ε, αλλά είναι βασική η πληροφόρηση, γιατί είναι βασική η πληροφόρηση, αλλά δεν μπορεί κανείς να τα διαβάσει όλα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο διάφανες είναι αυτές οι υποχρεώσεις πληροφόρησης μέσα στις νομικές διατάσεις για έναν μικρό έμπορο παραδείγματο χάρη που δεν τα καταλαβαίνουν μόνοι τους που χρειάζονται νομική συνδρομή και συμβουλή για να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν και να τα καταλάβουν. Στην καθημερινή πρακτική λοιπόν δεν είναι κάτι τέτοιο δυνατόν διότι βλέπω ε, από τους ε, ε, εμπόρους ότι για να πουλήσουν στο διαδίκτυο πρέπει να δημοσιεύσουν ορισμένες δεσμεύσεις ψηφιακά και πρέπει κανείς να εξασφαλίσει ότι υπάρχει αυτή η, αυτή η δυνατότητα γιατί δεν είναι προφανές για πολύ μικρές επιχειρήσεις και ε, περαιτέρω αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν και το ερώτημα είναι ε, τι, πόσο μπορεί να είναι το κόστος διότι βλέπουμε ότι στο γερμανικό δίκαιο ο, ο πολιτής έχει δικαίωμα είτε να ε, διορθώσει ε, και να επιδιορθώσει το προϊόν ή να προσφέρει ε, να το ανταλλάξει. Πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται εις ε, ε, ε, στο διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο και θα πρέπει ο έμπορος να μπορέσει να τα υπολογίσει στο κόστος του διότι θα είναι πιο εύκολο αν κάποιος του φέρει το προϊόν στο κατάστημά του να το επιδιορθώσει με μικρό κόστος ή να το αντικαταστήσει. Επίσης υπάρχει και το θέμα της παραγραφής το ένα θέμα είναι εάν χρειάζεται κανείς ε, ε, μία προθεσμία παραγραφής των απαιτήσεων στη δεκαετία, δηλαδή αν αγοράσω σήμερα ένα iPhone, ε, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Οπότε τα 10 χρόνια νομίζω ότι ξεπερούν κατά πολύ τον, τη διάρκεια ζωής αν όχι όλων των προϊόντων τουλάχιστον πολλών η πρόταση ε, από γερμαϊκή προοπτική θα έπρεπε να περιορίζεται σε διετή ε, διάρκεια της εγγύησης και ε, εκεί δημιουργούνται άλλα προβλήματα διότι τι θα γίνει τι θα γίνει τη, η απέτηση του πελάτη από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται αποζημίωση ε, και ο, ο πελάτης μπορεί να πει ότι χρειάζομαι μία προθεσμία εγγύησης από όταν το αντιληφθώ αλλά ο εμπόρος δεν είναι σε θέση να ξέρει ποια στιγμή αντελήφθη ε, ότι υπάρχει πρόβλημα ο αγοραστής του προϊόντος. Οπότε στην πρακτική ε, σαν έμπορος πρέπει να βασιστώ σε μία εγγύηση δεκαετίας και υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει καν προκύψει ακόμη στη συζήτηση. Πώς θα παρουσιαστούν τα στοιχεία αυτά σε έναν ισολογισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να καταρτήσουν ε, ε, ισολογισμούς και υπάρχουν προβλέψεις για ε, τέτοιες επιστροφές και αντικαταστάσεις και το πρόβλημα δημιουργείται λόγω του συνδυασμού του μη υποχρεωτικού δικαιώματος που πρέπει να εκπληρώνεται και να καλύπτεται και το, την εγγύηση της δεκαετίας. Οπότε ε, μας λέγουν ότι έτσι ε, δεκαπλασιάζεται ε, το, η δυνατότητα επιστροφών προϊόντων και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μεταφέρεται στους ισολογισμούς και μπορεί για ένα-δυο χρόνια ε, ένας, ε, ένας εμπορός να αποβεί Ε, Όσο, όσο περισσότερες επιστροφές υπάρχουν και όσες περισσότερες προβλέψεις ε, πρέπει κάποιος να έχει στον ισολογισμό του τόσο λιγότερα κέρδη υπάρχουν και αυτό δεν καλύπτει ε, την, ε, τον καταναλωτή και την προστασία του τουλάχιστον στο θέμα αυτό των εγγυήσεων και της παραγραφής των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων. Ε, λοιπόν στην αρχή. Εάν δεν μπορεί κανείς να καταρτήσει το CSL κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αποδεκτό και για τον έμπορο και για τον καταναλωτό, εάν δεν πιστέψουν και οι δύο, τουλάχιστον να πιστέψουν ότι είναι μια καλή επιλογή, τότε όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο το εγχείρημα ε, θα αποτύχει πριν καν ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι γιατί ε, καθυστέρησε πολύ η χρονομέτρηση σας, γι' αυτό και δεν είδατε καθόλου μέχρι το τέλος πόσος χρόνος είχε περάσει. Σας ευχαριστώ πάντως για τις παρουσιάσεις σας. Μας παρουσιάζετε το θέμα υπό διάφορα πρίσματα. Θα εμβαθύνουμε και στη συζήτηση. Έχουν έρθει και πολλοί συνάδελφοι εντωμεταξύ. Καλώς ορίζω τον κύριο Μπερλίνγκουερ από την Νομική Επιτροπή. Θερμό καλώς όρισμα κύριε Μπερλιγκουέρ. Ποιος ε, έχει απορίες ή θα ήθελε να θέσει ερωτήσεις ε, προς τους δύο καλεσμένους μας, την κυρία Κογιέν και τον κύριο Ζάιφερτ. Αν δεν θέλει κανείς ε, προς το παρόν να λάβει το λόγο, να ξεκινήσω εγώ με κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα της προστιθέμενης αξίας της νέας νομοθετικής πρότασης, ιδιαίτερα για τα ένομα βοηθήματα. Γιατί ακούσαμε ότι έχουμε πολύ πιο ισχυρά ένομα βοηθήματα στο κοινό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολίσεων, μα είπε ο κύριο ε, πρώτο μας ομιλητή, ενώ αμφισβήτησε αυτό το θέμα για το κατά πόσο είναι πρακτικά αυτά τα ένομα βοηθήματα ή αν θα τα δεχτούν ε, οι πάροχοι. Αυτό είναι ένα θέμα ισορροπίας που θα πρέπει να βρούμε. Οπότε ένα θέμα είναι αυτό, τα ένομα βοηθήματα και πώς όντως προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. Δεν ξέρω ποιο θα ήθελε να απαντήσει ή ποιο θα ήθελε να θέσει επιπλέον ερωτήσει. Η κυρία Σενάλοβα, αλλά πρώτα ο κύριο Βαμπ. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Φαμπ, αντιλαμβάνομαι για το, την... Ε, την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Ε, ε, όσον αφορά το iPhone που παρουσιάστηκε σαν παράδειγμα ε, ε, μπορούμε να αναρωτηθούμε για τις εγγυήσεις που προσφέρονται εάν θα υπήρχαν τα ίδια προβλήματα αν υπήρχε νέο ευρωπαϊκό δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες προσφορές από διάφορες πλευρές και τελικά φαίνεται ότι πολλοί εγκαταλείπουν την ε, ιδέα της ενιαίας αντιμετώπισης. Αλλά είπατε ότι είναι δύσκολο να βρεθεί μία μέση οδό ε, και ένα ενιαίο δίκαιο και νομίζω ότι στην περίπτωση Αλπενχόφτ που υποχρεώνεται ο ε, πολιτής να δεχθεί ε, το, δικαίωμα, το δίκαιο της χώρας στην οποία πουλάει ακόμη και αν δεν το γνωρίζει ε, δημιουργείται μια πολύ δύσκολη ε, κατάσταση και γι' αυτό νομίζω ότι από νομικής απόψεως χρειάζεται μια ενιαία νομική βάση. Με συγχωρείτε μια στιγμή να δω αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Κυρία Σενάλοβα, γιατί και εκείνη δήλωσε επιθυμία να θέσει κάποιες ερωτήσεις. Να ακούσουμε τις ερωτήσεις μαζί και μετά να δώσουμε το λόγο στους καλεσμένους για να απαντήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις στον καθηγητή Ζάιφερτ. Ε, και στην κυρία Κογέννη. Η κυρία Κογέννη είπε ότι φοβάται μήπως η θέσπιση του νέου καθεστώτος δημιουργήσει κάποιες ανισορροπίες στην αγορά ή περιπλέξει νομικά την κατάσταση και δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Ζάιφερτ, πιστεύετε μήπως ότι υπάρχει αντίφαση σε αυτά που μας είπε η κυρία Κογιέννη. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζάιφερτ γιατί περισσότερε ερωτήσει απευθύνθηκα σε εκείνον και μετά στην κυρία Γκογιέν. Και φυσικά θα περάσουμε και σε δεύτερο γύρο ερωταπαντήσεων. Ο κύριο Ζάιφερτ. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα που τέθηκε για την ε, ενιαία αντιμετώπιση βεβαίως ε, είναι πάντοτε χρήσιμο όταν υπάρχουν διασυνοριακές ε, συναλλαγές να υπάρχει ένα αξιόπιστο και κατανοϊκό δίκαιο με μία υποχρεωτική νομική βάση αλλά το πρόβλημα είναι το κόστος των συναλλαγών Λοιπόν, και μάλιστα ο φόβος του υψηλού κόστου των συναλλαγών διότι ε, ελέγχθη από ε, μία έρευνα του αρμοδίου επιμελητηρίου ότι 40-50% ε, επιχειρήσεων δεν θέλουν καν να προβούν σε διασυνοριακές πωλήσει γιατί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν οι πωλήσει 2.000 ευρώ δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει ότι θα φορτωθεί επιπλέον 10.000 ευρώ για τη μία συναλλαγή ε, τα οποία θα οφείλονται ε, σε, ε, σε περιπτώσεις των επιπλέον εξόδων για τη διασυνοριακή πώληση, εγγύηση κτλ. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι υπάρχει μία αρχή η οποία η οποία ε, είναι περιεργή δηλαδή μπορεί κανείς να επιλέξει ε, με, με, με ποιο σύστημα θα προβεί σε μια τέτοια εμπορική συναλλαγή ε, βλέπουμε όμως ότι είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει εξεταστεί επαρκώς και ενδέχεται να υπάρχει μια δυνατότητα επιλογής δικαίου που να μπορεί να γίνει υποχρεωτική και να προχωρήσει. Δεν όμως αυτό το θέμα μας σήμερα. Σήμερα είναι το CSSL, δηλαδή ένα προαιρετικό σύστημα. Δεν κατάλαβα όμως την ερώτησή σας και ίσως ε, θέλετε να την επαναλάβετε. Κυρία μου. Ναι. Ευχαριστώ, αλλά εν μέρη ήδη απαντήσατε στην απορία μου. Αυτό που ρώτησα ήταν ε, ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γκόγιαν. Ε, εντόπισε μια έλλειψη ασφάλεια δικαίου, κάτι που κατά τη γνώμη της θα επιβαρύνει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη προ προς αυτό. Πιστεύετε θα επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά νομίζω ότι σχεδόν απαντήσατε. Όντως, αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα. Και γι' αυτό γι' αυτό προσπαθούμε να καταρτήσουμε συστήματα σαν το CSL, ε, το θέμα της νομικής ανασφάλειας. Ένα νομικό πλαίσιο είτε είναι δεσμευτικό είτε είτε είναι προαιρετικό εάν δεν επιτύχει ε, την νομική ασφάλεια δεν θα επιβιώσει δεν έχει κανένα νόημα δεν μπορεί κανείς λοιπόν να εκπονήσει κάτι τέτοιο. Και πάντοτε ε, το θέμα στο οποίο επανέρχομαι είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για, τα, για τις Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ε, διότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει πάντοτε ο, ο κίνδυνος ότι θα επέμβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ανατρέψει την νομική βάση και τότε κανείς έμπορος δεν πρόκειται να δεχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Χρειάζεται μία ενιαία, αξιόπιστη και σταθερή νομική βάση ε, χωρίς ε, να σκεφτούμε ότι επιπλέον ο κάθε εθνικός νομοθέτης μπορεί να βάλει και το δικό του λιθαράκι. Και ουσιαστικά αυτός θα κάνει στο τέλος ό,τι θέλει. Από εκεί προέρχονται τα έξοδα των συναλλαγών, η δυσαρέσκεια και η απροθυμία μία να συμμετάσχει κανείς στο σύστημα και να παραδώσει προϊόντα. Οπότε υπάρχουν ορισμένα προϊόντα τα οποία μπορεί κανείς να αγοράσει μόνο στο εξωτερικό και όχι στη χώρα του. Μάλιστα. Τώρα θα σας δώσω το λόγο κύριε Αγκουγέν. Φαντάζομαι κύριο κύριος ο εισηγητής μας, θα γνωρίζει με ποιους τρόπους θα καταλήξουμε στη μέγιστη εναρμόνιση, γιατί ήταν, επαναλαμβάνω, συγκητή για την οδηγία τη προστασία του καταναλωτή. Δεν ξέρω, κύριε Κογιέν, έχετε κάποια σχόλια. Ναι, θα ήθελα να σχολιάσω τη δική σας ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, για την προστιθέμενη αξία αυτής της νομοθετικής πρότασης. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ε, των ένομων βοηθημάτων, αλλά όχι με προαιρετικό εργαλείο, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι καταναλωτέ χρήζουν καλύτερη προστασία και δικαιούνται καλύτερα με βοηθήματα, αλλά όχι με προαιρετικά μέτρα, γιατί είναι σαν να πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση ολοκληρώθηκε. Διαφωνούμε. Πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση έχει και μέλλον. Δεν περατώθηκε η διαδικασία αυτή. Πρόκειται για μια εξελικτική διαδικασία. Γίνεται προοδευτικά. Πριν από δύο χρόνια θα ήταν αδύνατο να καταλήξουμε σε συνένεση αλλά μπορεί μετά από τρία χρόνια να χρειαστεί να ξαναρχίσουμε και να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς και πολύ πιο ολοκληρωμένα ένομα συστήματα για να βελτιωθεί και η προστασία του καταναλωτή ακόμη περισσότερο. Είναι σημαντικό να κάνουμε τις αναλύσεις σταδιακά και προοδευτικά. Πάντως πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, αξίζουν ε, νομική, ε, ασφάλειες δικαίου και ενιαίας και ομοιόμορφης προστασίας παντού και όχι ένα προαιρετικό σύστημα που θα είναι παράλληλο με το εθνικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά το κόστος συναλλαγής, στην μελέτη επιπτώσεων έγιναν κάποιες προσωμιώσεις μόνο, πιθανολογήσεις ε, για το κόστος ε, για, την, για τις επιχειρήσεις ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών ε, για, από την εφαρμογή του νέου μέτρου. Τώρα θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος της αναζήτησης τέτοιων νομικών Ευρωπαϊκών συμβουλών για την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, Δικαίου Πολίσεων. Μάλιστα, ποιος άλλο θέλει το λόγο? Ο κύριος Βόρνερ και, και, ο κύριος Στανμάγερ μου φαίνεται είπε ότι θα ήθελε να μιλήσει. Σε λίγο θα του δώσω το λόγο. Ο κύριος Βόρνερ πρώτα όμως παρόλο που αργότερα θα λάβει το λόγο. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να κάνω ένα σύντομο σχόλιο απατώντας ε, στην ερώτηση που έγινε για το κόστος ε, συναλλαγών από ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή που υποτίθεται ότι υπόσχεται το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πωλήσεων. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το ισχύον νομικό καθεστώς προσφέρει κάποια νομική προστασία και δεν θα πρέπει το νέο καθεστώς να αυξάνει το κόστος συναλλαγής. Γιατί μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να προσφέρουν ένομα βοηθήματα που ξεπερνούν το, το δίκαιο. Ας μην υπερβάλλουμε λοιπόν. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιο, ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος για τη νέα ρύθμιση. Άλλωστε ε, σε μερικές χώρες μέλη η περίοδη παραγραφή είναι πολύ μεγαλύτερε από αυτέ που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Μερικέ φορέ ε, καλύπτουν όλη τη ε, ε, διάρκεια ζωή του προϊόντο. Οπότε τι θα γίνει με τη κατάσταση των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. Ενώ άλλες χώρες δεν έχουν καμία περίοδο παραγραφής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Θέλει ο κανείς το λόγο. Κύριε Στανμάγερ, πώς θα θέλετε να σχολιάσετε αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ευγενικό από μέρους σας που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν, η κυρία Κογέν επανειλημμένως τόνισε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούσουμε ως γνώμονα ε, ε, το κοινοτικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο. Μα έχουμε και τα δύο δίκαια ως γνώμονες. Το είπαμε από την αρχή ότι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο προστασίας του καταναλωτή που είναι τουλάχιστον τόσο υψηλό ε, ή και υψηλότερο από το κοινοτικό κεκτημένο, το ισχύον κοινοτικό κεκτημένο και είπαμε ότι σε σχέση με το εθνικό δίκαιο Γενικώ ε, έχουμε και συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας ή και υψηλότερο από τις εθνικές διατάξεις. Οπότε έχουμε διπλό γνώμονα, διπλό μέτρο σύγκρισης. Και χαίρομαι που ο καθηγητής ε, από το Βέλγιο είπε ότι κατά 99% το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί να προσφέρει ψηλότερο επίπεδο προστασίας. Τώρα, ε, ούτε είναι σωστό αυτό που είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαν να θεωρεί ότι έχει λήξει η εναρμόνιση. Λάθος, είπαμε και κατά την υποβολή της πρότασης ότι η πρόταση αυτή δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει καμία εναρμόνιση σε συναφείς ε, τομείς ή σε συγκεκριμένους τομείς. Και για το ψηφιακό θεματολόγιο, γιατί σε αυτό αναφερθήκατε, είπαμε εκεί, προβαίνουμε σε, μια εκτίμηση για να δούμε αν χρειάζονται και οι κανόνε εκεί κάποια εναρμόνιση. Πάντω, κανεί ουδέποτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είπε ότι δεν πρόκειται να υπέρθει περαιτέρω εναρμόνιση ή δεν επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση στο κοινοτικό κεκτημένο. Επειδή και γι' αυτό το λόγο θα προτείναμε το ΚΕΔ ω προαιρετικό. Επίση, συμφωνώ ότι το θέμα ε, για τις ε, μη καταχρηστικές συμβάσεις. Ναι, αλλά με ποια... Ε, ε συγγνώμη, για τα υποδείγματα συμβάσεων, για τις τυποποιημένε συμβάσεις. Ναι, αλλά με ποιο υπόδειγμα. Γιατί σε μερικέ περιπτώσει το κοινοτικό κεκτημένο προβλέπει μια ελάχιστη εναρμόνιση. Και δεν είμαστε, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ε, επειδή η διατάξη για, τον, για τους καταχρηστικούς λόγους είναι ελάχιστη εναρμόνιση. Κάποιος δικαστής δεν θα πει ότι η συγκεκριμένη ρήτρα ε, αντίκειται στο εθνικό δίκαιο για τους καταχρηστικούς ε, κανόνες. Αν έχουμε λοιπόν τυποποιημένε συμβάσει, υποδείγματα συμβάσεων, θα πρέπει να είμαστε ε, βέβαιοι σε ποια βάση συντάσσουμε αυτά τα υποδείγματα, με ποια βάση τα συντάσσουμε. Γιατί συνήθως έχουμε μοντέλα συμβάσεων με, ένα, με μία ενιαία βάση που είναι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο Πολίσεων. Τώρα, για το EDR και το ODR, αν είναι πραγματικός και ρεαλιστικός τρόπος ε, ε, για να προχωρήσουμε. Ακριβώς ένα μήνα μετά την πρόταση για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο Πολίσεων υποβάλαμε και μία πρόταση για το ODR και μία πρόταση για το ADR. Και μάλιστα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας και οι δύο προτάσεις και θα εγκριθούν ω ονούπο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι δύο προτάσεις αυτές σχεδόν κατατέθηκαν ταυτόχρονα, γιατί κατά τη γνώμη μας αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου ευρύτερου πακέτου. Ο κύριος Σάιφερτ μίλησε για την πληθώρα υποχρεώσεων ενημέρωσης. Όντως, θα πρέπει να αποφύγουμε κατακλυσμό των καταναλωτών από πληροφορίες. Αλλά όπως είπαμε και στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη, είδαμε ότι υιοθετήθηκε η υποχρέωση μια σειρά μιας σειράς πληροφοριών που απέβησαν πολύ χρήσιμες για τον καταναλωτή. Και μάλιστα έπρεπε ε, να πάρουμε από την οδηγία για το CRD όλες τις ε, υποχρεώσεις ε, για προ συμβατική ενημέρωση. Αλλιώς θα μπορούσε κανείς να παρακάμψει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου με το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Και αυτό και έπρεπε να περιλάβουμε όλες τις υποχρεώσεις προς συμβατική ενημέρωσης. Ό,τι αφορά το κόστος συναλλαγής για τους εμπόρους. Και είπατε ότι η εναρμόνιση εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους εμπόρους. Αυτό είναι εν μέρη σωστό και αληθές, γιατί η πλήρη εναρμόνιση, η πλήρης εναρμόνιση και όχι απλή εναρμόνιση, Όντω θα ε, καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα με ένα προαιρετικό εργαλείο όπως είναι το ΚΕΔ, αλλά το βασικό μειονέκτημα ε, αφορά τους εμπόρους που απευθύνονται μόνο στην εγχώρια αγορά, γιατί αλλιώ εξαιτία ε, της εναρμόνισης του νέου δικαίου θα υποστούν τεράστια επιβάρυνση, ενώ δεν θα έχουν κανένα αντισταθμιστικό πλεονέκτημα, γιατί τους άλλους δεν ενδιαφέρονται για διασυνοριακές συναλλαγές και απλώς θα αναλάβουν κάποιο κόστος χωρίς να έχουν κανένα κέρδος. Γι' αυτό και στη μελέτη επιπτώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι αυτή η προσέγγιση επιβάλλει κόστος μόνο στις επιχειρήσεις και στους εμπόρους που έχουν σε αντάλλαγμα κάποιες, κάνουν κάποιες οικονομίες από το διασυνοριακό κόστος συναλλαγής. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες. Καταρχήν, συμφωνήσαμε ότι σε περίπου 10 λεπτά θα ολοκληρώσουμε αυτό το δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης, οπότε έχουμε λίγο χρόνο ακόμη για κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις. Μου έστειλαν και ερωτήσει κάποιε οργανώσει καταναλωτών και εκπρόσωποι του. Για παράδειγμα, ε, ρώτησαν για την μελέτη επιπτώσεων και τις υποθέσεις της αξιολόγησης. Ίσως, κυρία Σενάλοβα και κύριε Μάγερ, σκόπιμο θα ήταν και για το ακροατήριο να μας επισημάνετε τις βασικές σας αμφιβολίες ως προς τη μελέτη επιπτώσεων, ποια κενά εντοπίσατε και τι ερωτήσεις έχετε συμπληρωματικές. Δεν ξέρω, όχι κατά τώρα αμέσω, αλλά κάποια στιγμή καλό θα ήταν να συμπληρωθούν και αυτά τα Κύριε ε, Μάιερ, έχετε ερωτήσεις προς τους ε, εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση στον κύριο Ζάιφερτ. Έχει σίγουρα δίκιο όταν λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν δυσκολίες και οι έμποροι να καταλάβουν περίπλοκη νομοθεσία και ανησυχούν για τη νομική βάση. Θέλουν μία ασφαλή νομική βάση. Θέλουν τώρα ένα εναλλακτικό σύστημα ε, εθελοντικό να μπορεί κανείς να επιλέξει σε ποιο δίκαιο θα βασιστούν, το μαθαίνουν, το διδάσκονται ε, και ε, ε, μπορούν στη συνέχεια να πούν ότι ναι, θεωρώ ότι αυτό το δίκαιο είναι ασφαλής νομική βάση για μένα ή διαφορετικά τι θεωρείτε ότι πρέπει να βελτιωθεί από τη σκοπιά του ε, μικρομεσαίου εμπόρου. Αυτό είναι μία ερώτηση η οποία δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με δύο λέξεις, διότι υπήρχαν διάφορα βασικά θέματα πρέπει να δει κανείς ε, τις διορθωτικές ε, λύσεις τα remedies την σειρά ακολουθίας της παροχής υπηρεσιών και ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτό όμως που εμένα με ενδιέφερε σχετικά με την αξιοπιστία μιας νομικής βάσεως είναι ακριβώς αυτά τα, αυτή η ακρογωνία λύθη, η, κατανο, η ευκολία κατανόησης για τον έμπορο όχι μόνο δηλαδή η κατανόηση από τον νομικό και τον ε, νομομαθή αλλά για τον έμπορο και ε, ε, στο, ε, στο εσωτερικό εμπόριο δεν μπορεί κανείς να εξοικονομήσει άλλα έξοδα της συναλλαγής αλλά μέσω του CSL και μέσω αυτής της οδηγίας πάντοτε δημιουργούνται ανάγκες νομικής πληροφόρησης και τουλάχιστον από τη δικιά μου πείρα πρέπει ο εμπορός να απευθυνθεί σε έναν νομικό, σε ένα νομομαθή οπότε αυξάνεται το κόστος ε, και αν είναι κάτι στιγμιαίο ίσως είναι λίγο αλλά διαφορετικά γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται αξιοπιστία σε διάφορα θέματα και ο χρήστης ο ίδιος πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβει τα βασικά σημεία αυτού του εχειρήματος και του νομικού κειμένου και ενδεχομένως αυτό είναι συγκεκριμένο πρόβλημα για τους Γερμανούς αλλά όταν θα υπάρξουν δεσμευτικές διατάξεις που θα ισχύσουν εις ε, την πρακτική τότε υπάρχει ένα πρόβλημα από πλευράς ανταγωνισμού δηλαδή εάν ε, οι ε, υποχρεώσεις πληροφόρησης δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα τότε ενδέχεται να δείτε, να λάβετε μία επιστολή η οποία θα σας κοστίσει 1000 ευρώ ότι από τις 97 υποχρεωτικές διατάξεις λείπουν από τις εξηγήσεις σας δύο. Είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο πρώτος μας ομιλητής, ο καθηγητής, καθηγητής Τόιν θέλει να προσθέσει κάτι. Ο κύριος Τόιν. Η κυρία Γκογιάν πρώτα και μετά ο κύριος Στέικ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι το επιπλέον ε, κόστος συναλλαγής ε, αφορά μόνο τους εμπόρους που έχουν διασυνοριακές συναλλαγές και όχι τους εμπόρου τη εγχώρια αγορά. Αυτή όμω δεν είναι προσέγγιση εσωτερική αγορά, γιατί στην ε, εσωτερική αγορά θα έπρεπε να έχουμε συνθήκε ίσου ανταγωνισμού. Και για τον καταναλωτή δεν ε, θα είναι ίδια η μεταχείριση αν πρόκειται ε, για σύμβαση με εγχώριο έμπορο και σύμβαση με επιχείρηση που έχει διασυνοριακές συναλλαγές. Εδώ υπάρχει επίση ε, μία σύγχυση, ενώ οι κανόνε τη αγορά θα πρέπει να προβλέπουν συνθήκες ε, ισότιμου ανταγωνισμού. Έχουμε μάλλον μέσω δηλαδή εργαλείο κατακαιρματισμού παρά εναρμόνιση στην περίπτωση του ΣΥΖΕΛ, του Κοινοευρωπαϊκού Δικαίου Πολίσεων. Ο κύριο Στάικ, για το ίδιο θέμα, ήθελα να πω μετά από αυτά που ακούσαμε και από τον κύριο Ζάιφερτ, ότι το κείμενο θα πρέπει να είναι κατανοητό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό όμω είναι κάπω ουτοπικό. Δεν νομίζω ότι ένα νομικό κείμενο μπορεί να είναι οδέποτε κατανοητό. Ούτε νομικοί μερικέ φορέ να η δικηγόροι δεν καταλαβαίνουν τα νομικά κείμενα. Φανταστείτε ο απλό άνθρωπο. Αλλά νομίζω ότι σε τέτοιε περιπτώσει μπορούμε να βρούμε μία απλούστατη λύση. Και αυτή τη λύση θα την προτείνουν οι, ε, ε, ε, οι δικηγόροι. Βέβαια, μερικέ φορέ για μικρές αξιώσει δεν χρειάζεται καν να καταφύγει κανεί στο νόμο, γιατί είναι δαπανηρή διαδικασία. Οπότε χρειαζόμαστε ένα σαφέ κείμενο στο ODR και το EDR. γιατί συνήθως ε, αποφασίζουν και επιλύουμε τις διαφορές με βάση την κοινή λογική μεταξύ λογικών και συνετών ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουν καλύτερα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τώρα για το κόστο συναλλαγή. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, γιατί υπάρχει ένα σύστημα που μπορούν να το επιλέξουν και με το ίδιο σύστημα να πραγματοποιούν τι συναλλαγέ του ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη για να μην αντιμετωπίζουν την κάθε ξεχωριστή τάξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντική μείωση στο κόστο συναλλαγή. Η μεγαλύτερη μπορεί να φανταστεί κανεί μάλιστα. Ευχαριστώ. Κανένα ε, μέχρι στιγμή δεν σχολίασε και ίσως πριν το αφήσουμε αυτό εκρεμέ. Ε, και να επανέλθουμε ίσως προς το τέλος ε, για κάτι που είπε η κυρία Γκόγιαν, κάποιες εναλλακτικές προτάσεις που έκανε. Ε, μίλησε για, τις, για τα υποδείγματα συμβάσεων, τις τυποποιημένες συμβάσεις. Βέβαια, ένα τέτοιο μοντέλο συμβάσεων, υπόδειγμα συμβάσεων, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και εύληπτο και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Και ναι, μεν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι πάντα εξοπλισμένε για να διαβάζουν και τα μικρά γράμματα των νομικών διατάξεων, αλλά ε, αν έχουν ένα υπόδειγμα συμβάσεων, ίσω το ε, καταλάβουν καλύτερα. Από την άψη διαφάνεια, νομίζω ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα το υπόδειγμα συμβάσεων. Επίση, όταν παρουσιάσουμε στους καταναλωτές και τους ε, εμπόρους το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων, θέλουμε να παρουσιάσουμε τον πυρήνα, τα κεντρικά σημεία και φυσικά τα πλεονεκτήματά του. Από το κείμενο τη ισχύουσα πρόταση ε, του κ. Σταμπερμάιερ, ίσω βελτιωθεί αργότερα, δεν είναι εμφανέ ίσω κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο τμήμα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μπερλιγκέρ θα έρθει το λόγο τώρα ή αργότερα, γιατί από ό,τι ξέρω είναι ο συνεισηγητής για το θέμα αυτό στη Νομική Επιτροπή. Οπότε είστε πρόσδεκτο στη συζήτηση, κύριε Μπελιγκόρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένο να θέσετε ερωτήσει, αλλά αν το επιθυμείτε, πολύ ευχαρίστω. Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο τμήμα της δημόσιας ακρόασης για ένα συγκεκριμένο τμήμα του κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου Αφορά ένα θέμα που αφορά και την προστασία για τα δικαιώματα του καταναλωτή και πρόκειται για το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένα ε, σημεία και πτυχές αυτού του δικαίου της υπαναχώρησης. Και ε, θα κάνουμε και μια σύντομη παρουσίαση του τι συμφωνήσαμε ε, με την άλλη επιτροπή για το health check. Αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα. Ο κύριος Κρίστοφερ Warner, που τον ακούσαμε και πριν από λίγο σε ένα σχολιασμό, είναι ε, νομικός εμπειρογνώμονας ε, της Βρετανικής Οργάνωσης Καταναλωτού. Παρακολούθησε αυτό το θέμα εκ του σύνεγγης και μάλιστα συμμετείχε και σε ομάδες εμπειρογνωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μας κάνει μια παρουσίαση για το σημείο αυτό. Και έχουμε και τον κύριο δόκτωρα Ρούπερτ Μπέρλινγχάουζεν που είναι εμπειρογνώμονας της Linklaters και θα μας παρουσιάσει το θέμα υπό το πρίσμα ενός ε, νομικού δικηγόρου και θα μας παρουσιάσει τις διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων των καταναλωτών και των απαιτήσεων των επιχειρήσεων για το θέμα αυτό του δικαιώματος της ε, υπαναχώρησης. Πρώτα ο κύριος Γόρνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σας μιλήσω για αυτό το θέμα σήμερα το απόγευμα. Μιλάω βέβαια εκ μέρους του WITCH Είμαι εκπρόσωπος της WITS, αλλά την ίδια άποψη έχουν και όλες οι οργανώσεις καταναλωτών ανά την Ευρώπη. Πολύ σύντομα λοιπόν. Τι είναι το WITS? Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση καταναλωτών στην Ευρώπη. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναξάρτητη. Αυτοχρηματοδοτούμενη οργάνωση που δεν βασίζεται ούτε σε επιχορηγήσεις από την κυβέρνηση, ούτε από χρηματοδότηση από μετόχους, ούτε από διαφημίσεις κτλ. Πριν έρθω τώρα στο θέμα της επαναχώρησης, θέλω να σας πω ότι συμφωνούμε και εμείς με τις ανησυχίες που ακούγονται για το ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για την προστασία του καταναλωτή. Και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι αυτό το μέσο που προτείνεται είναι και το καταλληλότερο. Γιατί θα επηρεάσει τα πράγματα και στο μέλλον. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που η Επιτροπή ΙΜΚΟ ασχολείται με το θέμα αυτό και βάζει και τα σωστά ερωτήματα ο καταναλωτής έχει να αποφεληθεί από κάτι τέτοιο. Και είναι και ερωτήσεις που θέτει και η οργάνωσή μας, το WITCH δηλαδή, ότι δηλαδή βελτιώνεται η ενιαία αγορά για τους καταναλωτές. Ακούσαμε ήδη διάφορα επιχειρήματα. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε να αποφελείται ο καταναλωτής. Ενώ εδώ με το νέο αυτό σύστημα που προτείνεται το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα πρόσθετο όφελος για τον ε, καταναλωτή. Το τελευταίο πριν περάσω στο δικαίωμα επαναχώρησης είναι ότι πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες του νέου αυτού συστήματος. Γιατί πιστεύουμε ότι παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και ερωτήματα αρχής μάλιστα πρέπει να καταλάβουμε κατά πόσο υπάρχει πραγματικά ανάγκη για ένα τέτοιο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων όπως προτείνεται. Τώρα, το δικαίωμα υπαραχώρησης φυσικά και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Και εδώ όμως πρέπει να απαντηθούν διάφορα ερωτήματα. Για να το συγκρίνω στην σχετική οδηγία με το ΚΕΔΠ, ξέρετε ότι το δικαίωμα αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο εφαρμόζεται σε περίπτωση εξαποστάσεως πωλήσεων. Και ο καταναλωτής έχει έτσι το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη για οποιοδήποτε λόγο και να επαναχωρήσει σε σχέση με τη σύμβαση που έχει συνάψει. Έχει 14 μέρες τη διαθεσή του από τη στιγμή που παραλαμβάνει τα αγαθά και έχει άλλες 14 μέρες για να επιστρέψει το προϊόν. Και ο έμπορος έχει 14 μέρες να του επιστρέψει τα χρήματά του. Και το, η σύμβαση θεωρείται ως να μην έχει υπάρξει ποτέ. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων τι προσθέτει σε όλα αυτά. Η οδηγία, όπως ξέρετε, εναρμονίζει το δικαίωμα αυτό επαναχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει να κάνει με τις συμβάσεις και τις εθνικές, εθνικό επίπεδο δηλαδή, αλλά και τις διασυνοριακές. Οπότε δεν βλέπουμε τι έχει να προσθέσει όλα αυτά το ΚΕΔΠ. Τίποτα, κατά τη γνώμη μας. Τα δικαιώματα που υπάρχουν για τον καταναλώτη είναι τα ίδια στις δύο περιπτώσεις. Εγώ δεν βλέπω να κερδίζει τίποτα ο καταναλωτής από την αρρύθμιση. Πολύ μικρές διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις ε, χώρες είναι θέμα διατύπωσης πιο πολύ. Εδώ όμως κινδυνεύει με το νέο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ε, σύγχυση. Σε μερικές περιπτώσεις πάντως θα υπάρξουν προβλήματα. Πρόβλημα ασφάλειας και βεβαιότητας. Εφόσον υπάρχει ένα σύστημα προαιρετικό. Η για ορισμένου καταναλωτέ, δηλαδή μπορεί να είναι πιο αδύναμο από ότι για άλλους το δικαίωμα αυτό. Και εδώ βλέπετε σε ποιες περιπτώσεις, σε ποιες χώρες δηλαδή ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές. Ακριβώς γιατί οι καταναλωτές είναι πολύ ευάλωτοι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρές, μικρής ε, αγαθά. Αν για παράδειγμα, ισχύσει το μέτρο αυτό, δεν ε, πλήττεται το δικαίωμα κάποιου ο οποίος έχει βάσει αυτή της ρύθμιση αγοράσει κάτι στη Γαλλία. Για περιπτώσεις που έχουμε συμβάσεις για αγαθά αξία κάτω των 50 ευρώ, το δικαίωμα αυτό χάνεται εντελώ με την ρύθμιση σε διάφορε χώρε, τι βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, και σε πολλέ άλλε χάνεται σε πολλέ περιπτώσει όταν πρόκειται για αγαθά αξία κάτω των 50 ευρώ. Εφόσον λοιπόν μοιάζουν τόσο πολύ τα δικαιώματα στις δύο περιπτώσεις, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο χρειάζεται νέα ρύθμιση. Και αφού μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις θα έχουμε μείωση των δικαιωμάτων. Ο καταναλωτής πώς θα μπορούσε να επιλέξει μόνο εμπόρους οι οποίοι δεν λειτουργούν κάτω από το νέο σύστημα αλλά χρησιμοποιούν το εθνικό δίκαιο. Μπορούνε. Δεν μπορούν και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην βρίσκουν και έμπορο ο οποίο να μην έχει επιλέξει το νέο σύστημα η μόνη επιλογή που έχει είναι να αγοράσει ή να μην αγοράσει καθόλου μερικές φορές. Αν έχει μονοπόλιο ο έμπορος, πώς ε, θα μπορέσει να βρει άλλη λύση ο καταναλωτής. Η επιλογή δηλαδή τελικά που έχει είναι να αγοράσει ή να μην αγοράσει το αγαθό. Και πείτε πώς θα ξέρει ο καταναλωτής τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο σύστημα του Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πολίσεων και την ε, οδηγία που ισχύει μέχρι τώρα. Δεν είναι οι έμποροι αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν τον καταναλωτή να καταλάβει περισσότερο τι ισχύει. Έτσι κι αλλιώς το FATSIT δεν δίνει λεπτομέρειες για να γνωρίζουν οι καταναλωτές σε λεπτομέρεια τα δικαιώματά τους. Αλλά είναι και θέμα αρχίσει. γιατί ο καταναλωτής θα έπρεπε να μπορεί να έχει την επιλογή επίσης ώρες και όχι έτσι όπως γίνεται εδώ. Ο στόχος μας είναι η προστασία του καταναλωτή, που είναι ο δύναμος κρίκος σε αυτήν τη συναλλαγή. δεν αιτιολογείται καθόλου η μείωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε αυτή την περίπτωση. Γιατί όπως είπαμε καλύπτονται εδώ πέρα μόνο οι πωλήσει εξ αποστάσεως. Το δικαίωμα λοιπόν αυτό υπαναχώρησης μπορεί να μοιάζει πολύ στις δύο περιπτώσεις, αλλά η διατύπωση όπως είπαμε και πριν διαφέρει που μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά το δικαίωμα αυτό καθ' αυτό, αλλά μπορεί να ερμηνευτεί η διαφορά. Και το άρθρο 4 του παραρτήματος 1 να ερμηνευτεί αυτόνομα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι πρόκειται για δύο παράλληλα καθεστώτα. Η οδηγία από τη μια και το κέδβα από την άλλη. Τίθεται θέμα αρχής, όπως ε, είπαμε και πριν, για τους ε, καταναλωτές μας. Πώς θα φροντίσουμε να υπάρξει μια συνεκτική συνέχεια που θα δώσουμε στην περίπτωση που έχουμε την ρύθμιση. Ποια είναι η λύση λοιπόν. Πρέπει να συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε κατά πόσο όντως ο καταναλωτής θα έχει κάποιο όφελος από τη νέα ρύθμιση και ας προσπαθήσουμε να βρούμε και άλλες μεθόδους που μπορεί να είναι προτιμότερες, όπως για παράδειγμα συμβάσεις ε, ε, μοντέλα, πρότυπα συμβάσεων ή έναν κώδικα διοντολογίας. Δεν θα πρέπει να στερήσουμε από τον καταναλωτή τα δικαιώματα που έχει μέχρι τώρα. και ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφεληθούν. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο μας. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed, also for keeping very much time. Σας ευχαριστώ θερμά και ιδιαίτερα σα ευχαριστώ που σεβαστήκατε για το χρόνο σα Και τέλος, τελευταία παρουσίαση από εμπειρογνώμονα πριν ε, περάσουμε και σε άλλες ερωτήσεις και απαντήσει. Δόκτωρ Ρούπερτ Μπέλιγχάουζεν, παρακαλώ έχετε 10 λεπτά. Äh, Ευχαριστώ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σήμερα μιλώ για την ενονόματι ε, του, συλλόγου, του δικηγορικού συλλόγου της Γερμανίας από τις ε, πλευράς της ε, ενός ε, γερμανού επαγγελματία στον τομέα. Διότι ε, πρέπει να καλύπτουμε ε, την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει νομολογία από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια αλλά επιπλέον και εμεί συμφωνούμε ότι ένα ενιαίο δίκαιο πολίσεων στην Ευρώπη όπου ο πολίτης θα μπορεί παντού να αγοράσει, αγοράσει τα εμπορεύματα με τον ίδιο τρόπο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για τις ε, μικρομεσές θα ήταν ε, μια θαυμάσια λύση. Το σημερινό θέμα μας ε, δεν μας αποκαλύπτει πολλά διότι το θέμα της υπαναχώρησης δημιουργεί προβλήματα και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα συγκρίσιμα. Έχω όμως να πω τα εξής επ' αυτού. Βλέπετε πάνω στην πρώτη διαφάνεια ότι το ευρωπαϊκό δικαίωμα πολίσεων όπως και τα 27 εθνικά σχετικά νομο... και 27 σχετικές νομοθεσίες προσπαθούν να εναρμονίσουν τουλάχιστον σε έναν κατώτατο παρανομαστεί. Δηλαδή ε, το δικαίωμα του καταναλωτή είναι παντού εξίσου σημαντικό, ε, δεν είναι όμως ο μόνος λόγος του ενιαίου ευρωπαϊκού δικαίου πολίσεως ούτε της ε, σχετικής νομικής τάξης εξού και δεν πρέπει εκ προημίου να ρωτήσουμε τι θα μας προσφέρει επιπλέον το ΣΥΣΛ ε, πέραν του εθνικού εμπορικού δικαίου αλλά πρέπει να δούμε τι ε, προσφέρει πέραν των δυνατοτήτων ε, και αυτό πέραν της στενής νομικής καλύψεως πρέπει να επιτρέψει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς όπως είπε και ο Βάλγος συνάδελφος, κατά τρόπον ώστε οι προδιαγραφές που θα ισχύουν ε, για την προστασία του καταναλωτού ε, παντού να ε, είναι δεδομένες μέσω του ΣΥΖΛ. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα του δικαιώματος υπαναχωρήσεως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ε, σαν παράδειγμα κατά τρόπον ώστε να δούμε τι αποτελεσματικό μπορεί να επιφέρει το ΣΥΣΛ διότι θα υπάρξει μία πλήρης εναρμόνιση και στο ε, δικαίωμα υπαναχώρησης αλλά στην ελάχιστη εναρμόνιση ε, θα έχουμε ένα κατακαιρματισμό διότι τα εθνικά ε, ε, οι εθνικές νομοθεσίες πολίσεως θα εφαρμόσουν αυτή τη διάταξη διαφορετικά πράγμα το οποίο δεν θα επιτρέψει μία πλήρη εναρμόνιση και αυτό το συζητήσαμε σήμερα σχετικά με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης του πολιτή και ε, ε, ακριβώς εδώ μπορεί ε, να αποδειχτεί η σημασία του ΣΥΖΛ διότι θα επιτρέψει ένα μπορικό δίκαιο νέο το οποίο δεν είναι επιβαρημένο και προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες παντού στην ίδια χρονική στιγμή για να προστατευτεί ο καταναλωτής και αυτό πρέπει να είναι ενδιαφέρον όχι μόνο για τον καταναλωτή αλλά και για τον επιχειρηματία. Αλλά ε, ε, πιστεύω ότι έτσι δεν θα υπάρχει κατακαιρματισμός και θα υπάρχει μία μεγαλύτερη εναρμόνιση των διαφορετικών νομοθεσιών στα 27 κράτη-μέρη. Γι' αυτό είναι βασικό το εγχείρημα αυτό και γι' αυτό ναι μεν καλύπτει τον καταναλωτή αλλά ξεπερνά το στόχο της οδηγίας προστασίας του καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε τι προσφέρει ε, εφόσον το δικαίωμα υπαναχώρησης ε, σε όλα τα κράτη ε, θα είναι ίσο εάν δεν μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής ένα προϊόν σε οποιαδήποτε χώρα ένα προϊόν διότι δεν την προσφέρει ο πολιτής ο οποίος φοβάται να προσφέρει ένα προϊόν σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά όπου υπάρχουν 27 διαφορετικές ε, νομοθεσίες ενώ στην Αμερική υπάρχει μία σχέση η οποία επιτρέπει να συνεργαστεί κανείς με τις 27 νομοθεσίες στην Ευρώπη ε, ενώ εμείς εδώ προς το παρόν πρέπει να έχουμε 27 διαφορετικές προϋποθέσεις θέσεις πωλήσεως ενώ στην Αμερική υπάρχει ένα ενιαίο κείμενο. Πρέπει να δούμε λοιπόν εάν το εγχείρημα αιτιολογεί το κόστος της προσπαθίας και βλέπουμε ότι ο πολίτης που μένει σε ένα μικρό κράτος μέλος δεν μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν διότι δεν προσφέρεται καν. Όταν λοιπόν υπάρχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης ε, και το ε, ε, θα περιοριστώ σε ε, λίγες μόνο παρατηρήσεις από την νομοθεσία προστασίας του καταναλωτού διότι βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν οι σχετικές ρήτρε που αναφέρονται στο δικαίωμα υπαναχώρησης και δεν καλύπτεται έτσι μόνο ο καταναλωτής αλλά συγχρόνως τα δικαιώματα και του επιχειρηματικού και το καταναλωτή και στις επόμενες σελίδες βλέπουμε ότι τεκμηριώνεται η ε, θέληση ε, του παρόχου των υπηρεσιών του πολιτή να εφαρμόσει το υψηλό επίπεδο της ε, παροχής υπηρεσιών βλέπουμε ότι ξεκινάμε με το δικαίωμα υπαναχώρησης, της εξαιρέσεις και μία γενική επισκόπηση η οποία δείχνει πώς θα εφαρμοστεί αυτό το δικαίωμα, ποιος είναι οι προθεσμίες υπαναχώρησης, η πλήρη εφαρμογή της υπαναχώρησης, τις υποχρεώσεις του εμπόρου και ε, του καταναλωτή μετά από μία υπαναχώρηση και τέλος φτάνουμε εις ε, τις ε, συνδεδεμένες συμβάσεις και βλέπουμε ότι εδώ εφαρμόζεται η οδηγία για τον καταναλωτή και να, να ρωτηθούμε τέλος αν είναι υποχρεωτικές αυτές οι διατάσεις. Γενικώ όμως μπορούμε να δούμε ότι ε, ο ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει χρησιμοποιήσει για τις δευτερεύουσες συμβάσεις ακριβώς την ίδια διατύπωση και ε, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ε, ε, για τον επιχειρηματία, ιδίως τον μικρό επιχειρηματία, να προσφέρει το εμπόρευμά του παντού στην Ευρώπη διότι ε, χρειάζεται μέσω του συστήματος αυτού μόνο ε, να ε, εφαρμόσει ένα ενιαίο σύνολο νομοθετικό και μπορεί να αγοράσει και ο καταναλωτής πολύ περισσότερα προϊόντα με μικρότερο κόστος αντί να χρειάζεται να θα σε 27 διαφορετικές νομοθεσίες. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι διαφάνειες και οι πίνακες. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκριτικές πληροφορίες και συγκριτική ανάλυση μεταξύ των εθνικών δικαίων, της ε, οδηγίας για το δικαιώματα του καταναλωτή και του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου πωλήσεων. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα τέτοιο εμπεριστατωμένο έγγραφο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων μας και θα περάσουμε σε γύρω σχολείων και ερωτήσεων ως προς το δεύτερο τμήμα της δημόσιας ακρόασης και μετά θα αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα από τη δημόσια ακρόαση και αν στη συζήτηση θέλουν να λάβουν μέρος και οι εμπειρογνώμονές μας, πολύ ευχαρίστως. Απλώς δηλώστε αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στο κατάλογο θέλει κανείς ε, να θέσει ερωτήσεις. Δεν βλέπω κανέναν. Θα υποβάλω λοιπόν εγώ μερικές. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα και περιστατωμένη ανάλυση από τον κύριο Μπέλιγχάουζερ ε, και νομίζω ότι ε, καταλάβαμε ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο Περιλύσεων και η οδηγία για, την, για τα δικαιώματα του καταναλωτή δίνουν κάπως παράλληλα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οπότε ανακύπτει το ευρύτερο ερώτημα που μας επαναφέρει στο αρχικό σχόλιο του κ. Στέικ, αλλά και στα επιχειρήματα του κ. Γόρνερ και της κ. Γκοϊέν και ίσως από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αν σημαντικά ουσιαστικά τμήματα του Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου Πολίσεων συμπίπτουν ουσιαστικά με την οδηγία για τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών που μόλις έχει συμπεριληφθεί στις εθνικές ένωμες δύο εναλλακτικέ υπάρχουν. Η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή στην ε, μετάθεσή τους, στη μετάθεσή της στην Εθνική Νομοθεσία θα ωφελήσει τους καταναλωτές χωρίς να είναι περίπλοκο νομοθετικό εργαλείο ή μήπως το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πωλήσεων είναι ένα ανώτερο και πιο αναβαθμισμένο πακέτο μέτρων και προστασίας, γιατί υπερβαίνει ακριβώς την ε, οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και πολύ ενδιαφέρον ε, ο πίνακας του δόκτωρα Berlinhaus που μας παρουσίασε ε, τη σύγκριση των δύο με τις 27 διαφορετικές ε, κατηγορίες και την ε, μη συναφή ή κάπως συνάρτητη εφαρμογή ε, της ε, εναρμονισμένης νομοθεσίας. Οπότε ρωτώ, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων θα δώσει απάντηση στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν σωστά το εναρμονισμένο δίκαιο με συγκροτημένο τρόπο και τελικά καταλήγουμε σε ένα κατακαιρματισμένο και πολλαπλό καθεστώς. Ή έχουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία ε, στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο και ένας προβληματισμός της συζήτησης. Όσο ο Δ. Μπέλιγχάουζερ θέλει να δώσει πρώτος απαντήσεις, τις απαντήσεις, συγγνώμη. Πείτε μας ε, ε, γιατί έχουμε σε έναν αρμονισμένο καθεστώς 27 27 διαφορετικά τμήματα. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η ισχύουσα κατάσταση η οποία αποτελεί ε, το σημείο εκκινήσεως για ελάχιστη εναρμόνιση ότι δεν υπάρχει μία ενιαία κατάσταση αλλά και η πλήρης εναρμόνιση έχει όρια, φτάνει στα όρια της και το είδαμε αυτό. Εάν λοιπόν διαπιστώσουμε πολιτικός ότι δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει περαιτέρω τουλάχιστον με θεαματική πρόοδο, τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ε, μια πολύ καλή διέξοδος και συγχρόνως θέλω να απαντήσω και στα δύο ερωτήματα που θέσατε στο τέλος. Ε, καταφατικά ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να βοηθήσει στην εναρμόνιση και κάλυψη των δικαιωμάτων του καταναλωτή διότι οριοθετεί το χώρο και δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μία νέα νομοθεσία η οποία οποία δεν ε, ε, υπήρχε ε, προηγουμένως και επιτρέπει ενιαία να δρομολογήσει την προστασία των καταναλωτών. Το τι προσφέρει στην εσωτερική αγορά για μένα είναι πολύ θετικό διότι οι μικρές επιχειρήσεις έτσι θα μπορέσουν να πουλούν σε ολόκληρη την Ευρώπη τα προϊόντα τους με χαμηλότερες τιμές. Οπότε θα απαντούσα καταφατικά και στα δύο ερωτήματα και εδώ βλέπω την προστιθέμενη αξία του συστήματος αυτού και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Να ακούσουμε τον κύριο Γόρνερ και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σβάπ. Συνεχίζοντας α, τα επιχειρήματα του κυρίου Μπελινχάουζεν και φτάνοντας στα άκρα. Αν είναι δύσκολο ε, μια νομοθεσία να την εφαρμόσουμε στις 27 χώρες μέλη, ε, φανταστείτε τι θα γίνει με ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων που θα πρέπει να το εφαρμόσει κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και ο καθένας ε, θα ερμηνεύει κατά το δοκούν τις ε, οδηγίες του ΚΕΔ. Πιστεύετε ότι έτσι θα μειωθεί ο κατακαιρματισμός. Δεύτερον, σωστά κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτού και τα κοινά σημεία με το ΚΕΔΠ. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, ταυτοσημείες στο περιεχόμενο, αλλά όχι στον τρόπο διατύπωσης. Από νομική άποψη λοιπόν αυτό θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει δυσκολίες. Δυσκολίες ερμηνευτικές για παράδειγμα. Γιατί μία παράγραφος ε, χωρισμένη σε δύο μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική νομική ερμηνεία παρόλο που στην ουσία μπορεί να είναι κάπως πανομοιό, να είναι πανομοιότυπα τα έγγραφα. Επίσης, φαίνεται το δικαίωμα υποναχώρηση στο ΚΕΔΠ είναι ε, πιο ισχυρό από ό,τι στην οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Έχουμε δηλαδή δύο νομικά καθεστώτα που ξεκινούν από το ίδιο σημείο αφετηρίας, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο ε, τα επόμενα 5-10 χρόνια. Και αυτό νομίζω θα δημιουργήσει προβλήματα και στις επιχειρήσεις αλλά και στους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος ΣΒΑΠ δήλωσε ότι θέλει να λάβει το λόγο. Δεν ξέρω αν άλλος κανείς θέλει να λάβει επίσης μέρος στη συζήτηση. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ αυτό ε, το σκέφτηκα και θα το ελέγξω λεπτομερώς και θα υποβάλω μια σχετική τροπολογία αλλά η συζήτηση κύριε Πρόεδρε δείχνει ότι το σύστημα δεν βρίσκεται ε, στη, στα τελευταία στάδια των λεπτομεριακών τελειοποιήσεων αλλά ότι υπάρχουν ουσιαστικά, ουσιαστικοί προβληματισμοί. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Ουντερχάουζεν Μπέλιγχάουζεν, διότι ε, είναι σαφές ότι ε, το να καταφεύγει κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι ίσως η λύση αλλά όπως είπατε και εσείς αν υπάρξει πλήρης εναρμόνιση θα είναι απαραίτητο και αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ε, αντιλαμβάνουμε λοιπόν αυτούς που κατακρίνουν αυτή την πρόταση διότι ε, ορισμένοι είπαν ότι, ε, είναι, ότι η εναρμόνιση δεν θα ήταν υποχρεωτικά θετικό όπως το είπε ο κύριος Σέιφερ και η κυρία Γκόγεντς. Εγώ είμαι πρόσφατος ευρωβουλευτής και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι πολύ πιο παλιοί στην πιάτσα εδώ και γνωρίζουν τις δομές της εσωτερικής αγοράς. Εδώ λέμε ότι είναι κάτι που δεν είναι ούτε αρκετά καλό και είναι υπερβολικά περίπλοκο, συγκεκριμένα το ΣΥΖΛ και έτσι ε, αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει κάποια κινητικότητα. Εάν λοιπόν ο κύριος Ζάιφερ για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εσείς για το δικηγορικό σύνολο και η κυρία Γκόγενς ε, ενωθούν μαζί μας και μας πούν ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία μέση οδό υπέρ των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, ξέρουμε ότι ε, όπου και να, όπως και να προχωρήσουμε σε εθνικό επίπεδο διαφέρει η κατάσταση από τη μια χώρα στην άλλη. Γι' αυτό και η μόνη εναλλακτική λύση που προσφέρει η συγκήτρια είναι να ρωτά θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Αλλά εάν εσείς συμπράξετε θα πρέπει να ε, οθήσετε προς μία εναρμόνιση και στις οργανώσεις που εκπροσωπείτε διότι ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς υποψίες ότι στο μέλλον θα το απορρίψουμε. Με συγχωρείτε που ίσως έκανα αυτή την παρατήρηση τώρα αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι, νομίζω ήταν πολύ σημαντικό αυτό το σημείο θα δω αν ε, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και μετά θα επανέλθω στους καλεσμένους που ίσως σχολιάσουν αυτά που είπε ο κύριος Φαπ. Υπάρχουν ερωτήσεις προς τους ε, εμπειρογνώμονές μας. Όχι, οπότε μπορούμε να περάσουμε σε μια ευρύτερη συζήτηση που οριοθέτησε ο κύριος Φαπ. Για το τι μελγενέστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη σχετική πρόταση. Ακούσαμε διστάμενες απόψεις, ένα ευρύ φάσμα θέσεων και είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε επιλογές με βάση το ρεαλισμό. Επανέρχομαι στον κύριο Σάιφερτ και στην πρώτη του διαφάνεια που λέει ότι η ιδέα ενό προαιρετικού κοινού ευρωπαϊκού δικαίου πωλήσεων θα λειτουργήσει μόνο, είναι τόσο ισορροπημένο και για τις δύο πλευρές και το θεωρούν ως καλή επιλογή και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Σήμερα το απόγευμα δεν είμαι βέβαιος ότι διανύσαμε πολύ δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, στη τελευταία μας φάση της συζήτησης, τα συμπεράσματα, να μας πούν οι εμπειρογνώμονες μας ποια είναι η γνώμη τους για το τι μελιγενέστε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Και Νομίζω ότι η προειδοποίηση του κυρίου Σάιφερτ ήταν πολύ εύλογη. Κανένα δεν είναι ικανοποιημένο με την πρόταση αυτή. Φαντάζομαι θα το σχολιάσει και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κανεί δεν είναι ικανοποιημένο με την πρόταση αυτή. ίσως θα πρέπει να διαρευνήσουμε εναλλακτικέ προτάσει, εναλλακτικέ λύσει. Και ένα άλλο ζήτημα που χρήζει διαλεύκανση είναι και το τι πόρου έχουμε στη διάθεσή μα. Η κυρία Γκόγιαν είπε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παρούσα κατάσταση με βάση τις οδηγίες, την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρω, κάτι που προποθέτει και πόρου. Και ο κύριο Φαπ είπε ότι δεν είναι ίσω η κατάλληλη στιγμή να επενδύσουμε, να ε, ενώσουμε όλου μα του πόρου σε ένα νέο ε, προαιρετικό εργαλείο που είναι αβέβαιη λειτουργικότητα. Ίσως καλύτερα θα να επικεντρωθούμε στη βελτίωση της οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή, να φροντίσουμε να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μετά σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να επανέλθουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να το σχολιάσει ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως αυτές είναι οι διάφορες εναλλακτικέ που ανέκυψαν στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο διαδοχικά στους εμπειρογνώμονες. Δύο λεπτό καθένας παρακαλώ Πείτε μας τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Στόικ και μετά θα ζητήσουμε και μια διαφώτιση από τους εισηγητές μας, τους δύο συνεισηγητές. Έχουμε και το health check, το διαγνωστικό έλεγχο και τη μελέτη επιπτώσεων αυτών των προτάσεων. Ο καθηγητής Στόικ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι μέλη γενέστε. Νομίζω ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πωλήσεων είναι ένα είδο πιλωτική πρόταση. Ε, δεν προεξοφλεί τίποτα ω προ τι μελλοντικέ εξελίξει του κοινοτικού κεκτημένου. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί περιορισμοί για το κατά πόσο είναι, δυνα... είναι εφικτή η πλήρη εναρμόνιση. Οπότε, για καμία διετία, καλό θα ήταν να αφήσουμε το θέμα τη πλήρου εναρμόνιση και να δοκιμάσουμε αυτή την πιλωτική πρόταση, το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Και ίσως υπάρξουν κάποια προβλήματα κατακαιρματισμού και εφαρμογή τη οδηγία για, για τα δικαιώματα του καταναλωτή ή και για το ΚΕΔΠΑ, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Έχουμε και διαφορετικά νομοσυστήματα, συστήματα, αλλά έχουμε και τα δικαστήρια. Και ο ενοποιητικό παράγοντα φυσικά θα ήταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και για τα δύο νομοθετικά πακέτα, και για το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων και για το κοινό κεκτημένο, την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Αλλά α δώσουμε μια ευκαιρία στο ΚΕΔΠ ας μην το θεωρήσουμε ως το ίστατο βήμα, στο το τελευταίο βήμα. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία να αποδείξει την αξία του. Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Let's give Sizzle a chance. Δηλαδή ας αφήσουμε ε, να δώσουμε μια ευκαιρία στο Sizzle να λειτουργήσει και τα προσόντα για τον καταναλωτή υπερβαίνουν κατά πολύ τα μειονεκτήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν σε κάποιο κράτος μέρος ή από την κατάσταση η οποία σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στο καταναλωτή. Ε, δηλαδή το μειονέκτημα απολίας της προστασίας του καταναλωτή ε, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το πλεονέκτημα της ε, προωθήσεως της ενιαίας αγοράς και ε, σε μία εικοσαετία δεν θα θυμάται πια κανείς την εθνική νομοθεσία και ε, το ΣΥΖΛ πλέον ε, θα έχει συμπιέσει και αντικαταστήσει τις εθνικές νομοθεσίες επί του θέματος. Ο κύριος Ζάιφερτ, θέλω να απαντήσω στην, στην ερώτηση του κυρίου Σβάμπ σε ορισμένα θέματα δεν θα καταλήξετε ποτέ σε ομοφωνία. Μπορεί να περάσουν 15-20 χρόνια και θα τσακώνεστε ακόμη. Και ίσως είναι καλό που υπάρχει τώρα μία γενική αντιμετώπιση ε, από υψηλό επίπεδο οπότε όπως είπε και ο κύριος Μπέλιγχάουζεν δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το σύστημα πολύ εκ των, ε, εκ εταίρων θα πρέπει ε, να μην προεξοφλήσουμε από το πώς δουλεύει το σύστημα εάν θα προχωρήσουμε ή όχι. Νομίζω ότι εάν έχουμε το ΣΥΣΛ σαν μια εναλλακτική δυνατότητα αφήστε το να δουλέψει, να περιμένουμε δύο-τρία χρόνια, να δούμε πώς λειτουργεί. Μπορεί να είναι καταστροφικό, μπορεί και όχι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περιοριστούμε στο κεκτημένο του καταναλωτή σε σύγκριση με το ΣΥΖΛ. Μιλάμε για νέα μέτρα, νέα μέσα και ε, πάντοτε θεωρεί κανείς ότι υπάρχει μία αντιπαλότητα μεταξύ του ΣΥΖΛ και του κεκτημένου, πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές. Σας ευχαριστώ όλα κύριε Κογέννης. Όσον αφορά την ευθύνη τώρα της έλλειψης εναρμόνισης σε διάφορα θέματα, υπάρχει ο μύθος ότι αυτά τα κενά θα καλυφθούν και ότι θα έχουμε με, το, με τη νέα αυτή πρόταση Ευρωπαϊκού Δικαίου για τις πωλήσει ένα ενιαίο σύστημα, μια εναρμόνιση χωρίς κενά. Δεν είναι αλήθεια όμως. Δεν είναι αλήθεια. Προς το παρόν υπάρχουν ένα σωρό ερωτήσεις που δεν πολύ ακούγονται, αλλά θα προκύψουν έτσι και τεθεί σε εφαρμογή ένα τέτοιο προαιρετικό μέτρο. Άσε που το προαιρετικό δεν είναι καθόλου καλή επιλογή για τους καταναλωτές. Εντάξει, μπορείτε να πείτε ότι είναι ε, πειραματικό. Όχι, δεν πρέπει να παίζουμε με τον καταναλωτή και σε βάρος του. Τώρα, ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μοντέλα συμβάσεων, βεβαίω να μιλήσουμε με τι επιχειρήσει, όπως λέει και ο κύριος Σουάμπ, να έχουμε ένα soft law, μη δεσμευτικό ε, δηλαδή δίκαιο, το οποίο να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Αν διαπραγματευτούμε για κάτι τέτοιο, τότε και γίνουν καλά διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να χρειαστεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο για τέτοιου του συμβάσεις. Ο κύριος Βορνάν, ευχαριστώ. Πώς πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα στις χώρες μέλη πριν εντοπίσουμε ανάγκη για παρετέρω μέτρα. δεν ε, έχουμε δώσει την ευκαιρία στην οδηγία αυτή να μας δείξει κατά πόσο φτάνει όχι. Η εναρμόνιση έχει να κάνει με τις συμβάσεις ε, εξ που είναι βέβαια και ένα στοιχείο κλειδί για την ενία αγορά. Ας Δούμε λοιπόν τι γίνεται με την οδηγία και όπου εντοπιστούν δυναμίες, είτε πρόκειται για την ψηφιακή ατζέντα, είτε πρόκειται για άλλα προβλήματα, εκεί να δουλέψουμε, να άρουμε ότι νομικά εμπόδια υπάρχουν, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας για παράδειγμα, ε, σήμα, εμπορικό σήμα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις αλλά να αναγνωρίσουμε ότι το κύριο εμπόδιο για τις διοσυνοριακές δραστηριότητες μια επιχείρηση είναι το κόστος, ότι πρέπει εφόσον εγκατασταθεί σε μια επιπλέον χώρα να καλύψει το κόστος της εγκατάστασης, των φορολογικών κλπ. κλπ. Το νέο δίκαιο, πως όπως προτείνεται, προτείνεται για να βοηθήσει τους καταναλωτές Θα τους βοηθήσει όμως, θα αλλάξει κάτι. Γιατί πάντα ό,τι κάνουμε είναι προ όφελο των καταναλωτών. Ή θέλουμε να είναι προ όφελο των καταναλωτών. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ο κύριο Σάνμαιρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαντάζομαι, θέλει και εκείνο να μα πει τη γνώμη του για το τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια. Και μετά οι δύο συνεισηγητέ για να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτή. Παρακαλώ λοιπόν. Εδώ μας ρώτησαν διάφορα πράγματα το κοινό. Θα μας βοηθούσε πολύ αν μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι προτιμάτε μια πλήρη ένα πλήρη και λεπτομερή ορισμό για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των ε, πωλήσεων. Σωστά, γιατί πολλοί από τις οργανώσεις των καταναλωτών με ρωτάνε. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε και να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς το μέλλον. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν για να απαντήσω στην ε, αρχική ερώτησή σας στείλαμε και προς εσάς και προς τα Εθνικά Κοινοβούλια δύο πίνακες. Το πρώτο ήταν ένας πίνακας ο οποίος συγκρίνει το ε, ευρωπαϊκό ε, δίκαιο των πολίσεων και το συγκρίνει με ε, το κεκτημένο και το, ο δεύτερος πίνακας αναφερόταν ε, στο ευρωπαϊκό δίκαιο σε σύγκριση με τον ίδιο τομέα που δεν έχει αναρμονιστεί σε εθνικό επίπεδο και αναφέρεται στο ίμιση του, δικαι... του δικαίου πολίσεων και το ίμιση των ε, κρατών. Ε, θα ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή ε, στις αρχές του επομένου έτους, αλλά είχαμε μία ερώτηση από την κυρία Γκέπχαρ και τον κύριο Μάγερ. Προσπαθούσαμε να απαντήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα κατά τρόπον ώστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το όλο σύστημα να μπορέσει να υποφεληθεί. Όσον αφορά τις συζήτηση σήμερα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να διαπιστώσουμε ότι εις ε, ε, ε, το δεύτερο μέρος όλοι οι ε, εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα δηλαδή ότι θα προτείνει η νέα νομοθεσία το ίδιο, την ίδια προστασία των καταναλωτών η οποία ισχύει και τώρα είναι και κάτι λοιπόν το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε υπάρχουν δύο βασικά θέματα του κυρίου Μόνη σχετικά με ε, τις διατάξεις, ε, τις δύο διατάξεις όπου έχουν ε, διακριτική ευχέρεια τα κράτη-μέλη. Καταρχήν το δικαίωμα να επέμβει υπέρ του καταναλωτή ένα κράτος μόνο δικαίωμα υπάρχει στη Γαλλία στα premises contracts. Οπότε ουσιαστικά στον τομέα αυτό πρόκειται για μία διάταξη σχεδόν επουσιώδη και το δεύτερο είναι το επίπεδο από το οποίο εφαρμόζεται ε, το κατόφλι. Ξεκινάμε από τα 50 ευρώ διότι έπρεπε να προβλέψουμε έναν ελάχιστο, ένα ελάχιστο σημείο εκκινήσεως ε, και ε, υπάρχουν κράτη τα οποία ξεκινούν πιο χαμηλά, υπάρχουν και κράτη όπου δεν υπάρχει κανένα ελάχιστο επίπεδο εκκινήσεως. Αλλά ήταν δύσκολο να τα συνδυάσουμε όλοι. Αυτό όμως που είναι βασικό μετά τη συζήτηση ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Το ερώτημα είναι τώρα πώς αξιολογούμε την όλη διαδικασία. Και είπε ο κύριος Ρόν από τη μία πλευρά ότι δεν υπάρχει θέμενη αξία και ο κύριος Μπέλιν Χάουσεν είναι, είπε ότι η προστιθέμενη αξία είναι η δυνατότητα επιλογής του καταναλωτού. Όταν κοιτάμε λοιπόν την προστιθέμενη αξία πρέπει να δούμε ποια είναι τα δικαιώματα τα ουσιαστικά όπου δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία και εμείς πάντοτε είπαμε ότι πήραμε αυτά τα οποία υπήρχαν ή στην ε, οδηγία για ε, την προστασία των καταναλωτών και το μεταφέραμε στη νέα αυτή νομοθεσία. Υπάρχουν όμως ε, τρεις μέθοδοι οι οποίες έχουν ε, πλήρως εναρμονιστεί καταρχήν οι πληροφορίες, το δικαίωμα επαναχώρησης και οι προθεσμίες και υπάρχουν 10 νέες διατάξεις που είναι θέμενη αξία και προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτούς. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε μόνο στα οικονομικά ωφέλη που ανέφερε ο κύριος Χάουσεν αλλά και σε την νομική προστασία του καταναλωτού. Και τώρα έρχομαι στα σχόλια που έγιναν στην ευρύτερη συζήτηση, δηλαδή τις εναλλακτικές δυνατότητες. Δεν είχα καταλάβει κατά καταρχήν ε, ή μάλλον δεν είναι κατανοητό τι εμείς προσπαθούμε να περάσουμε όσον αφορά το πρότυπο των συμβάσεων. Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο είναι μία ενία νομική βάση ε, βάση της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους αλλά πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως των συμβάσεων. Και αυτή είναι η ιδέα μας. Η ιδέα λέει ότι με τους ανδιαφερόμενους μαζί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνη της ε, προβαίνει σε αλλαγές των συμβάσεων που που θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και αν μια μικρή επιχείρηση ε, θέλει να επιλέξει το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο σαν βάση πολίσεως μπορεί να το επιλέξει και συγχρόνων μπορεί να επιλέξει από το διαδίκτυο το πρότυπο συμβόλαιο συναλλαγής ε, το οποίο ε, έχει γίνει αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη και αυτό ε, ισχύει και αυτό δεν ισχύει για συμβάσεις άλλες που μπορούν να προσφερθούν. Ενώ έτσι η μικρομεσαία επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει το δικό μας πρότυπο και θα έχει την διαβεβαίωση ότι η σύμβαση γίνεται, αναγνωρίζεται παντού. Όσον αφορά ε, το σύστημα που είπατε κύριε Πρόεδρε, βέβαια έχουμε υπόψη μας τους πόρους των οργανώσεων των καταναλωτών και θα κάνουμε ένα πρώτο workshop με τα κράτη-μέλη για να συζητήσουμε ε, πώς ε, η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί ενιαία. Είναι μια σημαντική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταλήγω τώρα στο συμπέρασμα που απαντώντας στο ευρύ ερώτημα υπάρχει και ο κύριος Μπελινχάουζεν και ο καθηγητής Στόικ και οι άλλοι ε, ε, εμπειρογνώμονες εξετάζουν μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία είναι προσυζήτησης που ε, προσφέρουν οικονομικά ωφέλη και στον πολιτή και στον αγοραστή και έχουν τη δυνατότητα ε, να αναβαθμίσουν την αξία της συναλλαγής και ε, καθιστούν ε, τον τύπο ε, προαιρετικό, δηλαδή μπορεί κανείς να επιλέξει ε, εάν θέλει να ακολουθήσει αυτή την λύση και εάν ε, κατά αυτόν τον τρόπο ο πολιτής και ο καταναλωτής θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις νέες διατάξεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλια σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συνεισηγητές μας, πρώτα στον κύριο Μάγερ και μετά στην κυρία Σενάλοβα. Ένα-δυο λεπτό καθένας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνοψίζοντας, Συνήθως ο, ο κάποιος έχει κάτι, ε, θέλει να το πουλήσει και λέει το, πληρώ, το πουλάω για 100 ευρώ και κάποιος συμφωνεί στην τιμή και αγοράζει και αυτό γίνεται σε κάθε χώρα καθημερινά για εκατομμύρια ευρώ και στις 99% των περιπτώσεων δεν υπάρχει κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Ενώ εδώ δημιουργούμε την εντύπωση ότι σε κάθε εμπορική σύμβαση υπάρχουν συνεχή προβλήματα. Δέστε καταρχήν τι και αν υπάρχουν διασυνοριακές δυσκολίες στις συναλλαγές αυτές θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να τις επιλύσουμε. Πάμε λοιπόν στο, ε, στο διαδίκτυο, αγοράζουμε ε, ένα προϊόν για 120 ευρώ και όταν υπάρχει η σύμβαση λέγεται ότι θα παραδοθεί στη Γερμανία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το αγοράσουμε αγοράσουμε οπουδήποτε ενώ μπορείτε να βάλετε ε, ένα όνομα άλλου αποδέκτη σε μία από 12 άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εξ αυτών θα δείτε στις 12 επιλογές οι 5 θα είναι αρνητικές γιατί οι πολιτές δεν θέλουν να πουλήσουν εκεί και, δεν ξέρουν, και αυτό διότι δεν ξέρουν εάν θα λάβουν τα χρήματά τους ή εάν θα χρειαστεί να το αντικαταστήσουν εάν είναι ελαττωματικό. Δεν είναι ε, θέμα της οδηγίας, είναι θέμα να λύσουμε το κακό, το πρόβλημα. Το ότι οι έμποροι θέλουν να προσφέρουν προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά με ε, εξασφάλιση. Σήμερα ε, θέλουμε να ενοποιήσουμε όλες τις νομοθεσίες αλλά έτσι έτσι δεν υπάρχει βεβαιότητα. Μπορεί μόνο να προσφερθεί εναλλακτικά ε, και μπορούμε να επιλέξουμε ε, για την προστασία του καταναλωτή διάφορες νομοθεσίες. Και μετά θα ρωτήσετε σε κάποιον ο οποίος πουλάει ένα προϊόν 120 ευρώ, ξέρετε αυτή την νομοθεσία και θα σας πει πρώτη φορά την ακούω στη ζωή μου. Και ε, βλέπει λοιπόν ίσως γρήγορα την λύση εάν ε, υπάρχουν ε, περιπτώσεις σε ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Όποιος σήμερα δεν είναι σε θέση να λύσει και να πουλήσει τα, τα προβλήματά του και να πουλήσει τα, τα προϊόντα του με το ισχύον καθεστώς καθεστώς εναλλακτικό σας προσφέρουμε ένα νέο νομικό σύστημα να δούμε αν θα λειτουργήσει και αν δεν λειτουργήσει τίποτα δεν χάσαμε διότι από την αρχή λέχθη ότι θα παραμείνουν οι άλλες νομοθεσίες δεν αλλάζει τίποτα δεν καταργείται τίποτα δεν καταστρέφουμε τίποτα απλώς θα τα προσφέρουμε μία επιπρόσθετη δυνατότητα για την συναλλαγή μεταξύ του πολιτή και του αγοραστή. Τίποτα τίποτα άλλο δεν συζητάμε. Εάν δεν λειτουργήσει ε, δεν χάσαμε και πολλά. Κόστος, όπως ελέγχθη, ε, θα γίνει συζήτηση με τα εθνικά ε, κοινοβούλια η συνάντηση το Δεκέμβριο θα προχωρήσει, ε, θα γίνει τον ε, Ιανουάριο μία αξιολόγηση των επιπτώσεων από την Νομική Επιτροπή όπου θα υπάρξει μία σχετική ακρόαση νομική με τις επιπρόσθετες ερωτήσεις της εισηγήτριας κυρίας Γκέπχα κατά τρόπον ώστε το Κοινοβούλιο να κάνει τη δική του αξιολόγηση των επιπτώσεων και να ελέγξει άλλη μια φορά το όλο θέμα. Αυτά όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη και νομίζω ότι κατά άλλα η σημερινή ακρόαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, διαφορετικές απόψεις, αλλά εάν ξεκινήσουμε από την προϋπόθεση ότι θέλουμε προστασία των καταναλωτών, ενιαία αγορά, θέλουμε να μπορούν να αγοράσουν οι αγοραστές και να πουλήσουν οι πολιτές, αυτό είναι το μέλημά μας, τότε πιστεύω ότι αυτό το ε, εναλλακτικό σύστημα μπορεί να ε, ισχύσει προερωτικά να δοκιμαστεί και να δούμε ε, εάν οι 20-30 οδηγίες που το διέπουν μπορούν να συνεχίσουν και ε, υπάρχει δυνατότητα της χρησιμοποιήσεως του ΣΥΣΛ, χρησιμοποιείται η δυνατότητα για πρότυπες συμβάσεις και αν δεν το επιλέξουμε ε, θα σκεφτούμε κάτι άλλο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη αυτή η σύναψη και μας παρουσίασες ε, και το μελλοντικό μας χρονοδιάγραμμα. Πολύ χρήσιμο. Κυρία Σαναλόβα. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην αρχή της συζήτησης. Και θα ήθελα στα συμπεράσματα αυτής της ακρόσης ε, να θίξω τα πιο κεντρικά σημεία. Επίσης, όπως επισημάνατε και εσείς, θέσαμε κάποιες ερωτήσεις ε, για κάποια κενά της μελέτης επιπτώσεων. Κάποιος μίλησε για ένα σύστημα που δεν ε, επιβαρύνεται από κανένα ιστορικό άχθος. Αν αυτό όμως το ιστορικό βάρος είναι ένα δεδομένο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή για κάθε κράτος μέλος, το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Έχουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις για το κόστος συναλλαγή και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και κάποια στοιχεία που περιλαμβάνει η μελέτη των επιπτώσεων. Θα σας αναφέρω αυτά τα στοιχεία η αναθεώρηση του health check ε, της μελέτης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ελέγξει το κατά πόσο η μελέτη επιπτώσεων στήριξε τους υπολογισμούς του κόστου συναλλαγής στις νομικές υποχρεώσεις ε, των επιχειρήσεων με βάση το κανονισμό Ρώμη 1 σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσουν ε, νομικές προσφυγές με βάση το άρθρο 6. Δεύτερη ερώτηση. Η μελέτη επιπτώσεων έλαβε υπόψη το γεγονό ότι ε, επιχειρήσει που πραγματοποιούν συνοριακέ συναλλαγέ ε, ε, επιλέγουν ε, τοπικούς ανάλογα με το με, την, με το δικό τους ε, ένομο σύστημα και δεν προσαρμόζονται στις ε, χώρες, με, στις χώρες Ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, του μοντέλου κόστου που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη επιπτώσεων. Επίσης, εξέτασε κάποια στοιχεία για το κατά πόσο ισοδύναμα τεστ του άρθρου 6 της Ρώμης 1 εφαρμόζονται εμπράκτος και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις. Και άλλη ερώτηση. Η οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, από ό,τι φαίνεται, δεν έληφθη υπόψη στη μελέτη επιπτώσεων του ΚΕΔ, παρόλο που προβλέπει πλήρη εναρμόνιση βαστικό στοιχείο για τι πολλέ εξ μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οπότε η επιθεώρηση θα πρέπει να εξακριβώσει το κατά πόσο η οδηγία ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή έχει επιφέρει επιπλέον, ε, επιπλέον κόστος ε, συναλλαγής και, και ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον τελικό υπολογισμό. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη επιπτώσεων ε, εξασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων του κοινοτικού και εκτιμένου για, το, για τα δικαιώματα του καταναλωτού, ιδιαίτερα αυτών της οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή τα, χρησιμο... τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ε, στη μελέτη επιπτώσεων προβλέπουν διαφάνεια και, ε, και προστασία του καταναλωτού από την, τοπική, από την εθνική του νομοθεσία υπό ορισμένε προϋποθέσεις. Τι γίνεται ε, για τις ε, επιπτώσεις στι ε, στις διασυνοριακές τη της Συμφωνίας για την προστασία του καταναλωτού σε περίπτωση συμβάσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη των επιπτώσεων. Ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους. Νομίζω ότι σας αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα γιατί ήταν πολύ αξιόλογη η δημόσια αυτή ακρόαση. Και επίσης ε, να ευχηθούμε και πάλι περαστικά και γρήγορη στην κυρία Γκέφχαρτ να ευχαριστήσουμε την κυρία Σενάλβα που την ε, αντικατέστησε επάξια, τον κύριο Μάγερ και τη Γραμματεία για την διοργάνωση και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή. Νομίζω ότι ήταν ε, πραγματικά υποδειγματική αυτή η δημοσιακρόση, κρόση, γιατί πραγματικά έφτασε σε βάθος σε πολλά θέματα. Συγκεντρώσαμε αρκετέ ενδείξει για το τι με και ποια θα είναι τα μεταγενέστερα βήματα. Μπορεί να μην φτάσαμε κατά ανάγκη σε συμφωνία, αλλά τουλάχιστον ε, μπορέσαμε και αντλήσαμε κάποια γενικά συμπεράσματα. Θα κάνουμε μια ολιγόλεπτη διακοπή προκειμένου να εκενωθεί η αίθουσα από δεν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και το επόμενο θέμα, παρόλο που σας διαβεβαιώ ότι και η έκθεση κύρια Μπάστος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Περιμένουμε λοιπόν να, ε, ε, να φύγουν από την αίθουσα όσοι και θα συνεχίσουμε με την έκθεση της κυρίας Μπάστος. So, ladies and gentlemen, I think we should make a start on our... Συνεχίζουμε. Και περνάμε στην εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών πάνω στις οποίες έχει δουλέψει η κυρία Μπάστος με τους σκιώδεις εισηγητές για την ε, έκθεσή της μετά τη δημοσίευση της Επιτροπής για τους 20 κύριους λόγους ανησυχίας των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Εμείς το ζητήσαμε μετά την έκθεση υγρές. Όλους μας ενδιαφέρει πολύ και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες επιτροπές οι οποίες θα συνεισφέρουν. Έξι επιτροπές συνολικά, από όσο ξέρω. Πολύ καλό σημάδι. Αυτό δείχνει ότι η απήχηση ήταν μεγάλη και στους άλλους συναδέλφους από άλλες επιτροπές. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μπάστος να μας εξηγήσει πού περίπου βρισκόμαστε και τις ε, συμβαστικές τροπολογίες πρέπει να τις έχετε όλες στα χέρια σας γιατί τις μοιράσαμε. Οι ακροατές θα μας πούν τη γνώμη τους. Ο κύριος Ρέπο εδώ έχει κρυφτεί, δεν τον βλέπω πολύ καλά, αλλά τον εντόπισα. Ε, για τον κύριο Ροσφόρ, Ρωμάντος, από ό,τι κατάλαβα. Η κυρία Ρούλη δεν είναι εδώ, η κυρία Μακλάρκιν είναι εδώ. Ο κύριος Ντεγιόν δεν είναι εδώ. Ωραία, έχουμε καλή εκπροσώπηση σχεδόν εισηγητών. Παρακαλώ κυρία Μπάστος, παρουσιάστε μας τις συμβαστικές αστροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως ε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω τον καρπό των διαπραγματεύσεων και των διαβουλεύσεων που είχαμε με τους και ηγητές προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβαστικές ε, τροπολογίες προσπαθώντας να συμπυκνώσουμε σε αυτές τις 82 τροπολογίες που, που κατατέθηκαν για την έκθεση. Μία έκθεση που εκφράζει τους βασικούς λόγους ανησυχίας των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Πρόκειται για ανησυχίες και προβληματισμό που έχουν τεράστια εμβέλεια. Αφορά τις δεξιότητες, τα προσόντα, τις συντάξεις, επιστροφή εξοδων υγείας, ψηφιακές αγορές, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ΦΠΑ, ε, παροχή ενέργειας, το κόστος ενέργειας, ε, λογαριασμούς ενέργειας, τεράστιοι ε, και πολύ αριθμοί λόγοι της ανησυχίας των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ενόψε σε 20 με στόχο να βρεθούν κάποιες απαντήσεις από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κενά που δικαιολογούν αυτό τον προβληματισμό και την ανησυχία. Υπάρχει ένα έλλειμμα πληροφόρησης, υπάρχει ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και υπάρχει και ένα νομοθετικό έλλειμμα γιατί δεν έχουμε πάντα κοινοτική κοινοτικές αρμοδιότητες για να ανταπεξέλθουμε στις υψηλές προσδοκίες των συμπολιτών μας. Η έκθεσή μου πρώτα απ' όλα τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει το θέμα της διακυβέρνησης είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες, τους καταναλωτές δηλαδή, αλλά και τις επιχειρήσεις. Όπως είπατε και εσείς, ε, πολλές ήταν οι επιτροπές που συνεργάστηκαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης και συνέταξαν πολύ χρήσιμες γνωμοδοτήσεις και πολύ μεστές και εμπεριστατωμένες σε σχέση με τους 20 αυτούς ε, βασικούς λόγους ανησυχία. Και οι γνωμοδοτήσεις αυτές περιλήφθηκαν και στην έκθεση που κατήρτισα εγώ. Οι τροπολογίες ενθυγραμμίζονται με την πρόταση για αδρές γραμμές και όχι για την υποβολή συγκεκριμένων λύσεων για τους 20 αυτούς λόγους ανησυχίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους και οδησηγητές για την αγαστή συνεργασία, το συναλλακτικό το διαλλακτικό πνεύμα και το μεγάλο πνεύμα συνεργασίας που επικράτησε στις συναντήσεις και που δημιούργησε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα στις διαπραγματεύσεις. Τελικά καταλήξαμε σε 15 συμβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν τις αρμοδιότητες και των υπόλοιπων ε, επιτροπών που συνεργάστηκαν μαζί μας προκειμένου να καταρτήσουμε πιο εμπλουτισμένο και πιο, σωσ... πιο εμπλουτισμένη και πιο σωστή την έκθεση. Από τις 15 τροπολογίες μόνο σε μία υπάρχει διαφωνία από τους πράσινους και την ΚΟΕ. Πρόκειται για τη συμβαστική τροπολογία 5 που αφορά τις νέες αγορές που διανοίγονται με βάση το ηλεκτρονικό εμπόριο και την εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς τη συμβαστική αυτή τροπολογία. Πριν από λίγο έστειλα στους συναδέλφους των δύο ομάδων που διαφωνούν μια νέα διατύπωση που τροποποιεί την αρχική συμβαστική τροπολογία με στόχο να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες μας. Περιμένω τώρα να μου πούν τη γνώμη τους οι πολιτικές ομάδες ως προς τη νέα αυτή εκδοχή της συμβαστικής τροπολογίας 5. Κατά του λοιπόν έχω δύο μόνο σχόλια. Καταρχήν, ως προς την τροπολογία 22 του συναδέλφου De Jong, που αφορά την διαγραφή emergence of. Οι δύο αυτές οι λέξεις, emergence of, αφορά τις ε, νέες επιχειρήσεις, την εμφάνιση των νέων επιχειρήσεων και όχι όλες τις επιχειρήσεις ε, ανευρέσεως εργασίας ή ε, γραφείων εργασίας που έχουν κάπως λιγότερο έντιμο ή και απατηλό όπως αναφέρει η τροπολογία χαρακτήρα. Επίσης ένα σχόλιο ως προς την τροπολογία 78 του κυρίου Κορέντε Κάμπος που καλεί το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν την κοινοτική νομοθεσία σε μια δοκιμή, σε ένα τεστ ηλεκτρονικού εμπορίου. Η διαφωνία μου αφορά την μετάφραση, γιατί η αγγλική μετάφραση δεν έχει νόημα. Το τεστ που λέει η αγγλική μετάφραση. Προτείνω λοιπόν το εξή. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει όλη την νέα ε, κοινοτική ρύθμιση σε, ένα, σε μία δοκιμή, σε έναν έλεγχο υπό το πρίσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, e-commerce test. Νομίζω ότι έτσι διορθώνεται το γλωσσικό πρόβλημα που δημιουργούσε η τροπολογία του κ. Κορέντε Κάμπος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για την ε, συμμετοχή τους, αλλά να ε, ευχαριστήσω θερμά και τους εμπειρογνώμενους και τους συνεργάτες μας που συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε το στόχο για μια απλή, συνεκτική δομή της έκθεσης και εύληπτη. Επικεντρωθήκαμε στους 20 κύριους λόγους ανησυχίας των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και αποφύγαμε έμνοια κάποιων νομοθετικών προτάσεων που ήταν εκρεμής. Δεν θέλαμε να επαναλάβουμε την έκκληση ε, για υποβολή προτάσεων εφόσον τις προτάσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί. Για παράδειγμα, ηλεκτρονική υπογραφή, δημόσιες συμβάσεις ή ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ άλλων. Επίσης, συμφωνούμε με τις έγκυρες και ε, καλές προτάσεις που βελτιώνουν την έκθεση στις συμβαστικές τροπολογίες καλύψαμε πολλά σημεία και των γνωμοδοτήσεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους ε, συντάκτες ε, των γνωμοδοτήσεων των ε, υπόλοιπων επιτροπών αλλά και τους σκιώδης ηγητές. Χάρη στη συνεργασία όλων καταλήξαμε στην υλοποίηση του στόχου ενός καλού, απλού, εύληπτου πονήματος μιας ευανάγνωστης και μεστής έκθεσης. Νομίζω ότι θα συμπέσει αυτή η έκθεση με την, επέτειο, την 20η επέτειο της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει φυσικά να δοθεί μια συνέχιση, ε, μια και θα περάσει η, οδηγή, η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου του Στρασβούργου. Αυτά και ευχαριστώ θερμά στους συναδέλφους που ε, συνέβαλαν στην υλοποίηση της συμφωνίας για τις 15 αυτές συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ και για τους συντονιστές. Είναι ένα περίπλοκο θέμα για όλους, αλλά υπάρχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Ρίπο τώρα, η κυρία Μακλάρκιν, κυρία Ρούλε, εσείς, όχι. Καλώς. Άλλος κανείς, κάμπος, ναι. Και ο κύριος Μάντης μου είπε θα ξαναρχόταν, ε. Θα δούμε. Εκεί η κυρία Μπαστός βέβαια. Κύριε Πρόεδρε. Ξέχασα να πω πριν ότι ο συνάδελφος Ροσφόρ ήταν πολύ συνεργάσιμος και πολύ πρόθυμος και διαθέσιμος. Μάλιστα, πέσει 7 δικές του τροπολογίες, 69, 70, 71, 72, 76, 78 και 79, κάτι που διευκόλυνε κατά πολύ το έργο μου. Ξέχασα προηγουμένως να επισημάνω αυτή την πολύ σημαντική συνθήκη. Ωραία, θα το επαναλάβουμε όταν έρθει. Παρακαλώ, κύριε Ρέπο. Παρακαλώ εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μπάστος για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μαζί, ετοιμάζοντας την τόσο σημαντική αυτή έκθεση. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα δεν χρειάζεται να αποσύρουμε τροπολογίες, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις συμβαστικές τροπολογίες της ε, εισηγήτριας. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε, δηλαδή θα δεχτούμε συμβαστικές τροπολογίες. Καλώς. Αδυνάλλεται κανείς, κυρία Ρούλε. Στηρίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες, μας ικανοποιούν. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί σας. Η κυρία Μακλάρκιν τώρα. Όλοι τέτοια λέμε σήμερα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε αυτό το θέμα και για την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί της. Υπέβαλα διάφορες τροπολογίες για να ενισχύσω το αρχικό κείμενο, την πρόθεση, για παράδειγμα, του συστήματος MI, για να βοηθάμε τον κόσμο, για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και γιατί δεν πρέπει να ρυθμίσουμε υπερβολικά. Ό,τι κάνουμε να είναι αναγκαίο και να είναι καλά στοχοθετημένο, να δίνει πρόσθετη αξία. Συνεπώς, με, με ενδιαφέρει ο στόχος της καλύτερης ρύθμισης. Οι δοκιμές θα πρέπει να εφαρμόζονται με σωστό τρόπο, να υπάρχει συνοχή. Και συμφωνώ με τις ευαστικές τροπολογίες. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά να μας ακούσει. Ευχαριστούμε, Λέω Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την συνάδελφο Ρέζινα Μπάστος για την εξαιρετική της δουλειά, όπως επισήμαναν και προλαλήσαντες, και να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί της και Εστενίζομαι και εγώ τη νέα διατύπωση για την τροπολογία 68. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί δίνουμε έμφαση και προτεραιότητα σε 20 τομείς ε, παρέμβαση στην εσωτερική αγορά. Και σε ό,τι αφορά την εκρεμή συμβαστική τροπολογία, την υπαριθμό 15, θα ήθελα να πω ότι ήταν κρίμα να διαγραφεί η πρόταση ε, υπό την δημιουργία ενός τυποποιημένου κανόνα για τις ε, ευρωπαϊκές συμβάσεις. Είναι πολύ καλή αυτή η αρχή και θα ήταν κρίμα να χαθεί στη σύμβαστική ε, τροπολογία. Βέβαια όλα εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις και στη διεξαγωγή τους είναι εξαιρετικά ικανή γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Ε, η αρμόδια εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έρθει πολλέ φορέ και παρακολούθησε από την αρχή τη συζήτηση στην Επιτροπή μα. Θα τη δώσω το λόγο αν θέλει να σχολιάσει κάτι. Oh, Παρακαλώ, αλλά το μικρόφωνο σα δεν δουλεύει. Α, τώρα εντάξει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια πάνω απ' όλα για τα όσα μας είπε, για το πώς μας βοήθησε. Για μας δεν έχει λήξει υπόθεση. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον κατάλογό μας για να συγκεντρώνουμε ιδέες από τον κόσμο. Μας έχετε υποδεχτεί πολύ θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε. Αυτό είχα μόνο να πω, τίποτα άλλο. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Αύριο θα ψηφίσουμε στις 10. Αλλά προηγουμένως, 9 με 10, θα δουλέψουμε για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Είναι όμως και κλεισμένο το θυρών. Οπότε όλοι μαζί θα τα ξαναπούμε στις 10 αύριο το πρωί. Υπάρχει και ένα νέο newsletter. Να ξέρετε, όποιος θέλει αντίγραφα και όποιος θέλει να γραφτεί, να παίρνει ηλεκτρονικά, να γραφτεί. Κυρία Μπάστο, σας ευχαριστούμε, όπως επίσης και όλους τους κοιόδες συζητητές. Και αύριο θα ψηφίσουμε. Ελπίζω στην Ολομέλεια να μας δοθεί ευκαιρία να έχουμε μια καλή συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε όλοι μαζί αύριο στις 10.